Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ελπίζω να ήταν ε, παραγωγική, επικοδομητική η χθεσινή συνεδρίαση. Για προφανείς λόγους κάποιοι Γερμανοί συνάδελφοι είναι ιδιαίτερα απασχολημένοι αυτή την περίοδο, γιατί δεν πρόκειται να πάμε στη Τζαμάικα, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Στο σημείο 7 έχουμε την σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με το Hong Kong 20 χρόνια μετά την παράδοσή του. Είναι παρόν ο Άλαν Σμίθ, ο εισηγητής. Άλαν, θέλεις το λόγο. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Είπατε ότι είναι απασχολημένοι οι Γερμανοί ευρωβουλευτέ, θα μπορούσαν και χειρότερα, θα μπορούσαν οι Βρετανοί ευρωβουλευτέ να είναι ιδιαίτερα απασχολημένοι. Πάντω, ευχαριστώ του συναδέλφου για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για την έκθεση αυτή. Θεωρώ ότι ε, είναι σημαντική ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταφέρει να καταγράψει πώ έχει κατάσταση στο Χονγκ Κόνγκ, ένα σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και το υπόλοιπο τη Κίνα. Νομίζω ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ισορροπημένη προσέγγιση. Έχουμε όπως ε, και η να πακολουθεί μια ενιαία και μοναδική πολιτική, έτσι και εμείς ενίο μέτωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σάμιελ καθώς επίσης και τη Γραμματεία και τους βοηθούς από την πολιτική μου ομάδα, αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες για τη συμβολή τους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε σήμερα την έκθεση αυτή. Εκεί είμαι στη και τυχόν περαιτέρω παρατηρήσει. Σα ευχαριστούμε, Άλαν Σμιθ, λέει ο πρόεδρο. Δεν νομίζω ότι θα πάρει κανεί άλλο το λόγο, έτσι δεν είναι. Βλέπουμε ότι η Γκουέ έχει ζητήσει ονομαστική κλίση για τις τροπολογίες 47 και 98. Ναι, και έχει αυτό περάσει στον κατάλογο ψηφοφοριών. Άρα μπορούμε να αρχίσουμε την ψηφοφορία. ξεκινήσουμε λοιπόν. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47 με νομαστική κλίση. Το έχει ζητήσει η Γκουε. Άρχτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 20 υπέρ, 22 κατά. Τροπολογία 48 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 48, άρτη ψηφοφορία. Καλημέρα, Γιώργο. Πέρας. 20 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 52, υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 52, άρχιτη ψηφοφορία. Νομίζω ότι απορρίπτεται πάντως, λέει ο πρόεδρος. Πέρας. Απορρίπτεται. Είναι σαφές το αποτέλεσμα. Περνάμε στην 53. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση και για την 53. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 26 κατά 18 υπέρ. Συμβαστική 6 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία παριθμών 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 61, άρχιτη ψηφοφορία. Ένα λεπτό, Μισελ. Περιμέναμε εσά. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται 26 κατά 19 υπέρ. 62 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Χωριστή ψηφοφορία έχει ζητήσει ο συγητής. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84 των Λάινεν και Πίτσουλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση μάλιστα. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 87. Πέρας. 24 υπέρ, 21 κατά. Η 87 λοιπόν εγκρίνεται και περνάμε στην 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 88. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 23 υπέρ, 24 κατά. Τροπολογία 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασική τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 95 παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 96. Άρτη ψηφοφορία. 49 στα που έχουν ψηφίσει. Πέρας. 29 κατά, 19 υπέρ. Περνάμε στην 97 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 98 μονομαστική κλίση, άρθρη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 99 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη α, τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καταπίπτει, σε συγγνώμη. Πάμε στην 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 6. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται, είναι σαφές το αποτέλεσμα. Περνάμε στην 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 9, άρτη ψηφοφορία.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 απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση και τροπολογία 35, άρθρη ψηφοφορία. Ένας ακόμα πρέπει να ψηφίσει. Πέρασε. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 39 του συγητή υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται, έτσι δεν είναι. Ηλεκτρονική επαλήθευση 39. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ετολογική αναφορά τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την έκθεση όπως τροποποιήθηκε, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. <clears throat> Και εγκρίνεται 45 υπέρ, 5 κατά, συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Πάμε τώρα στο σημείο 8, λέει ο Πρόεδρος. Γυναίκες, ισότητα των φίλων και κλιματική δικαιοσύνη. Πολύ καλή ερώτηση. Ο κύριος Παντζέρη, ο εισηγητής, είναι παρόν, μάλιστα εκεί. Ο κύριος Γκάλα ρωτούσε, κύριε Παντζέρη, τι είναι κλιματική δικαιοσύνη. Μήπως θέλετε να μας εξηγήσετε πρωτού συνεχίσουμε. Είναι η δέκατη φορά που το εξηγώ στον ε, Γκάλα και αυτός δεν καταλαβαίνει, δεν φταίω εγώ, λέει ο κύριος Παντζέρη. Okay, Michael, bist du mit der Antwort einverstanden? Michael, συμφωνείς εσύ με την απάντηση αυτή? So we come to... Πάμε λοιπόν ε, στην ψηφοφορία. Δεν θέλει ο κ. Παντζέρη να πει κάτι άλλο, όχι. Μάλιστα. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 Ποιο είναι το πρόβλημα, λέει ο πρόεδρος. Για πάμε στη συμβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτω. 70 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ την 70 άρχεται η ψηφοφορία πέρασε απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 69 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 69 παρακαλώ. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 6 υπέρ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 της, του συνόλου της εγγνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Και πέρας. Εγκρίθηκε 44 έναντι 5. Συγχαρητήρια στον κύριο Παντζέρη. Right. It's 9.30. Λοιπόν, είναι 9 και μισή. Και μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο. Όχι, πρέπει να περιμένουμε λίγα λεπτά, διότι ο πρέσβης δεν είναι ακόμα εδώ. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, we now come... Κυρίες ε, και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, την ενημέρωση για την 14η διάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Ινδία που διεξήθη στο Νέο Δελχή στις 6 Οκτωβρίου. Όπω θα θυμάστε, πολλέ φορέ έχουμε τονίσει την ανάγκη για βαθύτερε σχέσει ε, εντό του στρατηγικού πλαισίου που συστάθηκε το 2004 και πράγματι έχει επιστρέψει ένας δυναμισμός ε, στη σχέση μας από την Σύνοδο του Μαρτίου. Αυτό γιατί και η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατικές οντότητες στον κόσμο έχουν μια ιδιαίτερη ευθύνη για την διατηρήση της παγκοσμίας τάξης. Σήμερα θα ανταλλάξουμε απόψεις για την πρόοδο των ε, σχέσεών μας ε, στην διάσκεψη κορυφής που έλαβε χώρα, όπως είπα, στο Νέο Δελχή στις 6 ε, Οκτωβρίου. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζω την πρέσβυρα, την ε, κυρία Γκαϊτρή ακόμα, πρέσβυρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο και την κυρία Ιζαμπέλ Ντελέτρ της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, η οποία είναι υποδιευθύντρια για την ε, Νότια Ασία προτείνω να ξεκινήσετε εσείς, ε, κυρία Πρέσβυρα, και μετά θα δώσω τον λόγο και στην κυρία Λάτση και θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μακάλιστερ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ε, εξοχότατη, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας ενημερώσω για την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Πρώτα απ' όλα, ε, από αυτή είναι η πρώτη φορά να έρθω στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερος για το ότι υπερψηφίσατε το σχετικό ψήφισμα για τις σχέσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 13 Σεπτεμβρίου. Ήταν ε, ένα πολύ επικοδομητικό ψήφισμα τεκμηριωμένο, εάν μου επιτρέπετε, και νομίζω ότι πραγματικά έδωσε τον τόνο για τη Σύνοδο Κορυφής ε, της 6ης Οκτωβρίου. Είχα λοιπόν την ευκαιρία να συναντήσω μέλη της Επιτροπής ε, και να τους ευχαριστήσω προσωπικά, αλλά ε, δράτω με τις ευκαιρίες να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύ επικοδομητική αυτή συνεισφορά πριν από την συνάντηση των ηγετών μας. Η Σύνοδος Κορυφής, ε, που ήταν ε, μόνο ημέρη, κατάφερε να έχει πολλά θετικά σημεία. Οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου, ε, Τούσκ και Γιούνκερ, συνάντησαν ε, τους ηγέτες μας ε, πριν και μετά τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό. Είχαμε πολύ λεπτομερείς συνομιλίες ε, και εμείς στην Ινδία είχαν την άποψη και νομίζω ότι συμφωνεί εδώ πέρα και η Κομισιόν ότι είχαμε μια επιτυχημένη σύνοδο και καταφέραμε έτσι να επεκτείνουμε τον διάλογό μας και τις κοινέ μας ε, προσπάθειες ε, και αποφασίσαμε μέσω μιας κοινή δήλωσης 53 παραγράφων που καλύπτει ουσιαστικά όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας από το διάστημα και την πυρηνική συνεργασία για μη στρατιωτικούς σκοπούς μέχρι την απειλή της ε, τρομοκρατίας και της ε, ριζοσπαστικοποίησης. Βεβαίως το εμπόριο ήταν πολύ ψηλά και βεβαίως ε, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί και τους δύο. Και ακριβώς εδώ πέρα αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την, τα θέματα τα οποία συζητάμε και να συζητήσουμε κάποια ζητήματα ως στρατηγική εταίρη μεταξύ των οποίων και το εμπόριο. Στο εμπόριο αποφασίσαμε ότι αντί να το αφήσουμε σε μία σχέση αγοραστή και πολιτή, θα έπρεπε να προβλέψουμε τομείς όπου θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια διαταραχή στην αμφίπλευρη ροή του εμπορίου να προλάβουμε τέτοιες ε, διαταραχές όπως κάνουν οι στρατηγικοί εταίροι, να συζητάμε τα ζητήματα, να προετοιμαζόμαστε, να είμαστε έγκαιρα προετοιμασμένοι έτσι ώστε να μειωθούν ε, αυτές οι διαταραχές ή τα αποτελέσματά τους εάν τελικά συμβούν. Αμέσως μετά είχαμε κάποιες συναντήσεις με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είχαμε, έναν... Είχαμε αρκετές αντιπροσωπείες που πήγαν στην Ινδία και συνεχίστηκε βεβαίως η δουλειά που κάνουμε και ήδη προγραμματίζουμε να εργαστούμε στην στρατηγική συνεργασία μας και το ότι θα επιτύχουμε πριν την επόμενη σύνοδο κορυφής που μάλλον θα γίνει στις Βρυξέλλες και άρα την αναμένουμε. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργό μας μετέφερε στους ηγέτε, τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την προτεραιότητα που αποδίδει η Ινδία στις ε, σχέσεις της και την στρατηγική συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίω ε, θεωρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σημαντικό πυλώνα σταθερότητας σε έναν κόσμο που αλλάζει, ε, σε έναν πολυπολικό κόσμο και μια δημοκρατία η οποία έχει τις ίδιες αξίες ε, στις οποίες αποδίδουμε και εμείς μεγάλη σημασία, όπως ο πλουραλισμός, ε, ο πολυπολιτισμός και ένα σύστημα διαφανούς διακυβέρνησης και κράτους δικαίου και αυτή τη στιγμή όπου έχουμε τόσες αλλαγές ε, στο σενάριο αυτό. Ε, αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και ο Πρωθυπουργός ε, μετέφερε στους Προέδρους ε, Συμβουλίου και Κομισιόν το ότι εμείς θεωρούμε την συνεργασία μας ε, αμοιβαίως επωφελή και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος μας. Η Ινδία έχει βεβαίως συμφέρον ε, στο να επιτύχει το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε κάθε λόγο να το στηρίζουμε. Επίσης, ο κ. Πρωθυπουργό είπε ότι οι σύνοδοι κορυφής ε, θα έδιναν τον τόνο για την ενίσχυση της ε, σχέσης. Επίσης ε, υπάρχει η παράγραφος 53 της κοινή δήλωσης και αν υπάρχει κάποια πτυχή που θα θέλατε να συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ ε, για να μην ο άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Πρέσβη. Κύριε Ντελάτρε τώρα, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς ε, σας ζητώ συγγνώμη γιατί ε, η διευθύντριά μας δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Την αντικαθιστώ λοιπόν Αντικαθιστώ την κυρία Καρολίν Βινό, που είναι η επικεφαλής για τον τομέα αυτό που καλύπτει και την Ινδία. Βρίσκεται στον Μπαγκλαντές όμως σήμερα, όπου συνοδεύει την κυρία Μογκερίνη. Ξέρετε ότι η κυρία Μογκερίνη μετέβη στον Μπαγκλαντές από την Κυριακή. Σας ζητώ λοιπόν συγγνώμη για αυτή την αλλαγή τελευταία στιγμής. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ, που κάθομαι δίπλα σας κυρία Πρέσβη. Θα ήθελα προφανώς να επιβεβαιώσω τα όσα είπατε όσον αφορά την αξιολόγηση της, του πολυθετικού πνεύματος που είχε αυτή η Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας που όντως είναι μια σύνοδος που ατένισε περισσότερο το μέλλον και που διεξήχθη σε απλές μιας καταπληκτικής ατμόσφαιρας. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια πιο σταθερή βάση για τη στρατηγική μας συνεργασία και έχουμε πλέον και μια συγκλίνουσα προσέγγιση όσον αφορά τις μελλοντικέ προκλήσεις. Όντως, ο Πρωθυπουργό της Ινδίας είπε ότι έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος και καλωσόρισε την προδραστική προσέγγιση που έχουμε πλέον στα πλαίσια της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ινδία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνοδος λοιπόν ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και θετική, οδήγησε συγκεκριμένα αποτέλεσμα, όπως είπε και η πρέσβης. Έχουμε ένα μακροσκελές κείμενο, το οποίο συνοψίζει τα συμπεράσματα της συνόδου αυτής και καλύπτουμε πάρα πολλά ζητήματα, ζητήματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας και συμφωνήσαμε επί ε, τριών επιπλέον δηλώσεων για την καταπολέμηση τρομοκρατίας, για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, για την πρόθεση της καθαρής ενέργειας και για την ε, ευφύ και βιώσιμη αστικοποίηση. Συμφωνήθηκε επίση ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η συνεργασία μα σε ζητήματα ασφάλεια, ιδίω όσον αφορά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία κοινό μέλημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας, αλλά και στο ζήτημα της κυβερνοασφάλειας, καθώς επίσης και στο ζήτημα του φοπλισμού, της μη μετάδοσης πυρηνικών όπλων και της ασφάλειας στη θάλασσα. Είπαμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, ριζοπαστικοποίηση που λαμβάνει η χώρα στο διαδίκτυο. Είπαμε επίσης ότι θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε πολυμερές επίπεδο στα πλαίσια του GCTF, του Παγκοσμίου Φόρουμ για την καταπολέμηση της Χρηματοδότερησης της τρομοκρατίας. Είπαμε επίσης ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιες προκλήσεις, ανθρώπινα δικαιώματα, μη διάδοση πυρηνικών όπλων, μετανάστευση, κλιματικές αλλαγές, G20, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και οι μεταρρυθμίσεις επίσης που θα πρέπει να γίνουν. Όσον αφορά τι εξωτερικές σχέσεις, την εξωτερική πολιτική. Αυτό μας απασχόλησε κυρίω κατά τη διάρκεια του γεύματο εργασία. Καλέψαμε περιοχές και χώρες όπως το Νεπάλ, το Μπαγκλαντέ, το, Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, καθώς επίσης και την Αφρική, την Τουρκία και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Είπαμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας όσον αφορά το Αφγανιστάν και την Αφρική. Όσον αφορά τώρα το εμπόριο, εμπόριο και επενδύσεις, ε, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ε, σε ένα κοινό δρόμο πρόοδου ότι θα πρέπει να καταβληθούν εκ νέου προσπάθειες προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, για, την για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Στα πλαίσια της υπουργικής διάσκεψης του Μαρακές του ΠΟΕ ασχοληθήκαμε με το ζήτημα αυτό και οι διαπραγματευτέ για την συμφωνία αυτή ελεύθερων συναλλαγών συναντήθηκαν ήδη την προηγούμενη εβδομάδα στο Νέο Δελχή. Τώρα, όσον αφορά τι απαιτήσει διατροφική ασφάλεια, ασχοληθήκαμε με το ρύζι μπασμάτι. Οι ανησυχίε πάντω καλύφθηκαν στα πλαίσια μια πολύ επικοδομητική συζήτηση και θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά την πρέσβη, η οποία πραγματικά συνέβαλε πάρα πολύ επικοδομητικά στο να επιληθεί το, το πρόβλημα το οποίο είχε προκύψει. Συμφωνήσαμε για μια δέσμη ε, αντισταθμιστικών μέτρων που προασπίζουν τα, συμφέρα, τα συμφέροντα των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον ε, σχετικό κανονισμό της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε να κάνει με τις εισαγωγές Ριζιού μπασμάτη. Δεν καταφέραμε όμως ακόμα να καταφέρουμε να πείσουμε την Ινδία να δημιουργήσει έναν ε, οικονομικό διάλογο υψηλού επίπεδου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εξακολουθούμε και πιστεύουμε, όπως είπατε και εσείς κυρία Πρέσβη, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε παράγοντες που αναστατώνουν την ομαλή ροή του εμπορίου. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει εκ νέου να υποβάλουμε μια πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να έχουμε αυτόν τον οικονομικό διάλογο υψηλού επίπεδου, στα πλαίσια του οποίου θα μπορούσαμε να καλύψουμε επίση και επενδύσει εποφελείς και για τι δύο πλευρέ και θα μπορούσαμε να δούμε ποια άλλα βήματα μπορούμε να καλύψουμε για να προωθήσουμε περισσότερο το διάλογο αυτό. Όσον αφορά τώρα τι τρει επιμέρου δηλώσει. Ξέρετε ότι ε, όσον αφορά την καθαρή ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές, προωθούμε την άποψή μας ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρω συμφωνία των Παρισίων και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί συνεργασία σε πάρα πολλού ε, τομεί. Συμπεριλαμβανομένων και εδώ πέρα γίνονται λίγο πιο τεχνικές οι παρεμβάσει μου. Αποθήκευση ενέργεια, ε, ηλεκτρική κινητικότητα και ανανόσιμε πηγέ ενέργεια μεταξύ άλλων. Η Ινδία είναι μακροχρόνιος εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετώπιση των κλιματικών αλλαγών και πρόσφατα έγινε και μία συνάντηση στο περιθώριο ε, μιας συνόδου που είχαμε με τον Καναδά προκειμένου να προωθήσουμε τα ζητήματα αυτά αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Τώρα η συνεργασία όσον αφορά την International Solar Alliance και εκεί θέλουμε να βαθύνουμε περισσότερο τη συνεργασία μας και θέλουμε να θεσπίσουμε μια καλύτερη πλατφόρμα συνεργασίας. Μολονότι ε, δεν συμμετείχατε στην ε, προηγούμενη εκδήλωση, φαντάζομαι ότι τουλάχιστον θα συμμετάσχετε στην επόμενη. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δημιουργήσει και έναν ε, επίσημο διάλογο για τις κλιματικές αλλαγές με την Ινδία. Συμφωνεί και η Ινδική πλευρά, επομένως θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την πρόταση αυτή. Τώρα, η κοινή δήλωση για την εταιρική σχέση όσον αφορά την ευφύ και βιώσιμη αστικοποίηση. Έχουμε θέσει πάλι εδώ προτεραιότητε και στόχου προκειμένου να έχουμε μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά την ανάπτυξη των πόλεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει αναλάβει πολύ σημαντική δράση στον τομέα αυτό και προσπαθεί να εμπλέξει όλο και περισσότερες πόλεις και αρμόδιες αρχές στις πόλεις της Ινδίας, προκειμένου να συμμετάσχουν και αυτές περισσότερο σε αυτό το οποίο ονομάζουμε ολοκληρωμένη αστική διαχείριση. Θέλουμε επίσης να καταφέρουμε να διχειριστούμε καλύτερα κάποιες βασικές δημόσιες αστικές υπηρεσίες όπως διαχείριση των λιμάτων, ίδρυυση και το καθεξής. Και μάλιστα καταφέραμε να εγκρίνουμε την πρώτη χρηματοδότηση 500 εκατομμύρια ευρώ για το μετρό της ε, στην Μπαγκαλόρ και θα αρχίσει από, έχει ήδη αρχίσει από το 2016 να χρηματοδοτεί το μέτρο αυτό. Είπαμε ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να ενισχύσουν την ε, συνεργασία τους προκειμένου να υπάρχει μία συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, ερευνητικών ιδρυμάτων από την Ινδία. Υπεγράφει λοιπόν μια σχετική συμφωνία στο περιθώριο της προηγούμενης συνόδου προκειμένου ερευνητές ε, ταλαντούχοι από την Ινδία να μπορούν να επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε επίσης ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει μια πρωτοβουλία 30 εκατομμυρίων κοινή όσον αφορά το ζήτημα του νερού. Τώρα για την αεροπορία η Ινδία ανακοίνωσε ότι πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να θέσει σε επιχειρηματική φάση το, την οριζόντια συμφωνία επί αεροπορίας που υπογράφει το 2008, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Ινδία αναγνωρίζει πλέον τις αποφάσεις που έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργεί ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού όσον αφορά το τομέα της αεροπορίας. Αναφερθήκαμε επίσης στις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλει η Ινδία σχετικά με αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως όσον αφορά το κοινό θεματολόγιο για την κινητικότητα και τη μετανάστευση που υπεγράφει στη Σύνοδο του 2016. Η Ινδία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το σύστημα της μπλε κάρτας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος είπαμε ότι ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ινδικού Κοινοβουλίου και θεωρούμε, και αυτό λέγεται ήδη και στην έκθεση, ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τις πολιτικές και κοινοβουλευτικές μας σχέσεις με την Ινδία και να προωθήσουμε μάλιστα και ανταλλαγές μεταξύ αντιπροσωπιών των δύο κοινοβουλίων, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δύο κοινοβουλίων, των δύο βουλών της Ινδίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κρίστιαν Ταπρέντα, τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεσή του, την οποία επέβαλε σχετικά με την Ινδία. Και επίση είχαμε και θετικέ εξελίξεις από το τέλος τη Συνόδου μέχρι σήμερα στα πλαίσια του προγράμματος εργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018 που προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών μας με την Ινδία και πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε εργασίε για μια κοινή, ε, μια κοινή ανακοίνωση όσον αφορά την περαιτέρω στρατηγική μας ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας που θα υπογραφεί το 2018 αυτό αποτελεί μια ανταπόκριση στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση και Ινδία. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και προσβλέπω σε μια περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων μαζί σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Ντενάτχα, ευχαριστούμε την πρέσβη. Έχουμε περί την μισή ώρα, συνάδελφοι, για συζήτηση. Παρακαλώ, να μας υποδείξετε αν θέλετε να παρεμβέτε. Έχουμε τρία αιτήματα, Πρέντα, Φανόρτιν, Μπούχνα μέχρι στιγμής. Κανείς άλλος? Επομένως, ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Πρίντα και μετά τον κύριο Φανόρτιν. Προσπαθήστε να είσαστε να περιοριστείτε στα 5 με 6 λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Πρέσβη που βρίσκεται εδώ. Καταρχάς να χαιρετήσω αυτή την ευκαιρία που έχουμε για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα του, της 14ης Συνόδου, διάσκεψης μάλλον, του Οκτωβρίου, η οποία ήταν πολύ σημαντική και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας προς την ενεργοποίηση της ε, στρατηγικής εταιρικής ε, σχέσεως μετά από τέσσερα χρόνια σιγής. Και όπως όλοι οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν, Είμαστε απολύτω υπέρ τη ενίσχυση αυτή τη εταιρική σχέση ε, με σημαντικό όφελο και για τι δύο πλευρέ. Τώρα, η διάσκεψη αυτή κορυφή ήταν ένα σημαντικό βήμα προ την κατεύθυνση τη ενίσχυση αυτή και εγώ ήμουν πολύ ικανοποιημένο που είδα ότι η πτυχή της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ήταν στην καρδιά των συζητήσεων του Νεοδελχή. Όπως επίσης σχετικά με το γεγονό ότι διάφορα εδάφια της κοινή δηλώσεως αφορούσαν στο θέμα αυτό, όπως και στην καταπολέμηση τρομοκρατίας, δηλαδή θεματικές που είχαμε επεσκευαστεί στη γνωμοδότησή μας από τον ε, Σεπτέμβριο, με ικανοποίηση είδα ότι βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Τώρα, θα ήθελα να υποβάλω κάποια ερωτήματα στους ε, καλεσμένους μας. Καθότι και αυτοί συμμερίζονται την απόψή μου ότι ήταν θετικό το αποτέλεσμα της διάσκευσης. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τι θα θεωρούσε εκείνη ένα βήμα προς τα εμπρός ακόμα πιο αποφασιστικό. Δηλαδή τι θα θέλατε να δείτε μεταξύ των συμπερασμάτων που δεν το βλέπετε ως προσδοκία ένθεν κακήθεν, δηλαδή Ινδία και η ΕΔ. Αν δηλαδή εκπληρώσαμε το επίπεδο της φιλοδοξίας που είχαμε θέσει. Τώρα για την ε, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, η κυρία Μάλστρομ με την συνομολόγη της το συζήτησαν θα μπορούσε να ελπίσει κανείς να δει κάτι σαν φύλλο πορείας επί τη συνέχεια των συζητήσεων αυτών. Είμαστε κοντά σε ένα τέτοιο οδικό χάρτη ή θα συνεχίσουμε με κάποιες επαφές, με κάποιες ε, συναντήσεις οι οποίες δεν προχωρούν επί της ουσίας ίσως. Και τρίτο ερώτημα, ιδιαίτερα προς την κυρία Πρέσβη, επί της ε, τωρινής κρίσεως για τους Ροχίνγκια και γενικά για τις σχέσεις μεταξύ Μπαγκλαντές και Μιανμάρ. Εσείς θεωρείτε ότι επί τη βάση των συμπερασμάτων της διασκέψεως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία θα μπορούσαν να συντονίσουν τη θέση τους. Για παράδειγμα, ίσως ό,τι αφορά στην ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά επίσης σχετικά με την επίλυση, την πολιτική λύση που θα μπορούσε να βρει κανείς στο ζήτημα αυτό, το πρόβλημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος Τζέφρι Φανόρτιν, παρακαλώ. I don't know speak French. was amazing. Uh, Απίστευτο που μίλησε ο συνάδελφος γαλλικά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω την κυρία Κούμαρ, την κυρία Πρέσβη. Νομίζω ότι ακολουθεί τα λαμπρά βήματα των προκατόχων της και επιπλέον ε, έχει δεσμευτεί απολύτως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επεδίωξε και συνάντησε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετείχε στις συναντήσεις της Συνδικής Αντιπροσωπείας, την συνεδρίαση που είχαμε διοργανώσει για τις οικονομικές μας σχέσεις με την Ινδία. Γιορτάσαμε τον Τιβάλι μαζί και έχουμε και το Δημοκρατικό Φόρουμ της Νότιας Ασίας το απόγευμα στην Α1H1 οπου θα μιλήσει πάλι η πρέσβης μεταξύ άλλων διακεκριμένων ομιλητών για το όλο θέμα της Νότιας Ασίας την περιοχή αυτή που είναι σταυροδρόμη. Εκτιμώ λοιπόν την παρουσία της και την συμμετοχή της και τη δέσμευσή της με τις εργασίες και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι η Ινδία θα έπρεπε να είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στρατηγικούς εταίρους για τα ευρωπαϊκά έθνη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πάντοτε μένει λιγάκι στο περιθώριο. Μιλήσαμε για το εμπόριο, μιλήσαμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την αντιμετώπιση της πειρατείας, τα κοινά συμφέροντα και αξίες που έχουμε το ενδιαφέρον μας σε μελλοντικές ε, τεχνολογίες, σε βιώσιμη ενέργεια, καθαρό νερό, την καταπολέμηση των νόσων, πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Και τι σημαντική χώρα υπερδύναμη θα είναι η Ινδία. Η οικονομία της είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ασία ε, έχουμε ευρύτατο πεδίο δραστηριότητας και συνεργασίας είναι προφανές. Συμμετείχαμε και εμείς σε συναντήσεις της Ινδικής Αντιπροσωπείας στην ε, Ινδία και συναντηθήκαμε με υπουργούς ε, και πολλούς άλλους διακεκριμένους ομιλητές οι οποίοι πάντοτε μας καλωσόριζαν θερμά. Επισκεφτήκαμε επίσης την ειδική βιομηχανία, φορείς της οικονομίας, στην Μπαγκαλόρ και αλλού, αεροναυπηγική, όλη αυτή η πολύ σημαντική κλάδη της οικονομίας και τα κοινά πεδία δραστηριότητας που μπορούμε να έχουμε. Μιλήσαμε για την ε, διάσκεψη κορυφής και τα αποτελέσματά της, τα πορίσματα και νομίζω ότι αξίζει να υπογραμμίσει κανείς ε, την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα τη συνεισφορά των 500 εκατομμυρίων στο έργο του μετρό της Μπαγκαλόρ. Το ανακοινωθέν ήταν 10 σελίδες και 53 εδάφια. Ε, πραγματικά θα ήταν πολύ καλύτερα να ήταν δύο σελίδες. Με κάποια βασικά πολιτικά μηνύματα. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές συνεργασίας, αλλά αυτές τις οποίες επανερχόμεθα είναι οι διμερείς σχέσεις, οι εμπορικές και οι επενδυτικές. Εγώ προσωπικά δεν κατανοώ γιατί, για ποιο λόγο δεν προοδεύουμε πιο αποφασιστικά. Το 2007 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις και όπως και οι πρέσβεις και εγώ έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, η διατύπωση του ανακοινοθέντος είναι περίπου να λέμε ότι πρέπει να συζητήσουμε ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δηλαδή είναι κάπως ανεπαρκές και για τις δύο πλευρές. Και διερωτώ δεν υπάρχει επαρκής βούληση εκατέρωθεν για να προχωρήσουμε σε μια πλήρη συμφωνία. Είμαστε μήπως υπερβολικά φιλόδοξοι. Μήπως θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο επιφυλακτικοί με μια λιγότερο φιλόδοξη συμφωνία, μια τομεακή, κάποιες τομεακές συμφωνίες, πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε απτά και συγκεκριμένα. Ε, κυρία Πρέσβη, είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι από την παρουσία σας και την δραστηριότητά σας και τη συμμετοχή στις συναντήσεις αυτές. Νομίζω ότι μπορούμε πάρα πολλά περισσότερα να κάνουμε. Ο κύριος Μόντι είναι ένας πολύ δυναμικός Πρωθυπουργό έχει κινητοποιήσει τη χώρα και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δράξουμε τις ευκαιρίες που μας ανοίγονται πιο αποφασιστικά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Τζέφρι. Τώρα έχουμε τρεις συναδέλφους που θέλουν τον λόγο. Ο κύριους Φράιν, Τάνοκ και Μπούχνα. Κάποιος άλλος. Προτείνω λοιπόν να δώσουμε στην πρέσβυρα και την κυρία Ντέατρη από 5 λεπτά, οπότε 3 λεπτά ο καθομελητής. Ξεκινάμε τον κύριο Φρόιντ. Σας ευχαριστώ. Θα σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και Πρέσβη, θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να γνωρίζω, μια που το θέμα της κλιματικής αλλαγής δεν προέκυψε στην αρχική σας ε, δήλωση, αναρωτιέμαι πόσο συζητήθηκε αυτό το ζήτημα, ειδικά υπό το φως πρόσφατων ιστοριών για την ρήπανση στην Ινδία που έχει ε, λάβει φοβερές ε, διαστάσεις ε, και δεν περιορίζεται πλέον. Ειδικά υπό το φως του γεγονότος ότι από ό,τι φαίνεται η Ινδία σε αντίθεση με την Κίνα δεν αναζητά τόσο πολύ εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή δεν ακούμε κάτι τέτοιο. Και τι είδους ε, συνεργασία βλέπετε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα που βεβαίως ε, θα αποτελούσε έναν ενδιαφέροντα εταίρο για το ζήτημα της ε, κλιματικής αλλαγής, γιατί μιλάμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα ζητήματα που ανέφερε ο κύριος Φανόρντεν, αλλά Εάν δεν ελέγξουμε την κλιματική αλλαγή, τίποτα από όλα αυτά τελικά δεν θα γίνει. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε λίγα περισσότερα για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Τάνοκ κατόπιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω και να συγχαρώ την κυρία Κουμάρ που είχα την ευκαιρία να συναντήσω στο Στρασβούργο πριν από λίγους μήνες όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της. Πριν από 18 χρόνια ήμουν ένας εκ των ιδρυτών της ομάδας φίλων της Ινδίας πριν ε, το Κοινοβούλιο ε, αποκτήσει αντιπροσωπεία. Οπότε μετά η ομάδα μας ε, κατέστη περιττή. Αλλά από την πρώτη στιγμή λοιπόν Ήμουν πολύ ενεργός στο θέμα. Και θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση που αφορά την Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων που σέρνεται δυστυχώς εδώ και καιρό. Γράφει ο τύπος ότι ένα από τα προβλήματα ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο ε, δηλαδή όσον αφορά το αίτημα Mode 4 του ΠΟΕ για έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θεωρήσεων ειδικών λογισμικού από την Ινδία για να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό ήταν ένα από τα ζητήματα που μπλοκάρισε τις διαπραγματεύσεις και βεβαίως από την άλλη πλευρά υπήρχε ο φόβος για τις ε, Βρετανικές υπηρεσίες, ε, τις νομικές και τις τραπεζικές για το πώς θα διεισδύσουν στην ειδική αγορά που αυτή τη στιγμή προστατεύεται. Σημαίνει αυτό λοιπόν ότι το Brexit το 2019 θα βελτιώσει τις ε, πιθανότητες ε, να συνάψουν επιτυχώς μια συμφωνία ελευθερεμπορίου ή e 27. Σας ευχαριστώ και Τάνοκ και τέλος ο κύριος Μπούχνερ. Κύριε Πρέσβη, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που δέχεστε τις ερωτήσεις μας. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη. Επί 30 έτη ήμουν καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο στην Γερμανία και σε αυτή την 30 έτη πορεία δεν ε, είχα δει κάποιον Ινδό φοιτητή σε υψηλό επίπεδο, αυτό το οποίο λέμε σήμερα μεταπτυχιακό. Και αντιστρόφως, όταν, όταν μιλάμε για Γερμανούς στην Ινδία, επίσης δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Ε, δεν το αναφέρω επικριτικά, απλά εμείς ε, δεν βλέπουμε Ινδούς ε, φοιτητές. Μπορεί να βελτιωθεί αυτό. Δεύτερον, σε κάποιες εβδομάδες θα πάω στην 11η Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες και άκουσα ότι η παλιά Ινδική πρόταση ε, που αφορά τελικά το να επιτραπούν τα μεγάλα αποθέματα τροφίμων θα φύγει ξανά το τραπέζι. Ε, τι σημαίνει αυτό, θα μας στηρίξει τελικά η Ινδία θα παραμείνει σταθερή, θα αντισταθεί σε αυτές τις τάσεις κάποιων μεγάλων χωρών για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Δεν ε, βλέπω άλλα σχόλια από εσάς. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, έχω μία σύντομη ερώτηση. Κυρία Πρέσβη, με συγχωρείτε. Ελπίζω όλοι να θέλουμε να διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός ε, ε, διακοινοβουλευτικών επαφών μετά την επίσκεψη του Προέδρου του Ινδικού Κοινοβουλίου σε εμά, αλλά βεβαίως και την επίσκεψη της δικής μας της αντιπροσωπείας ε, στο Δελχή. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι εάν υπάρχει κάποια σχέδιο να επισκεφθεί η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ινδικού Κοινοβουλίου της Βρυξέλλες. Ε, σας έχουμε ήδη απευθύνει πρόσκληση ε, όταν ήμασταν στο Δελχή. Λοιπόν, ξεκινήστε εσείς και μετά θα ακούσουμε την... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας ξεκινήσω με το δικό σας το ερώτημα. Προφανώς ε, είμαστε υπέρ των ε, ανταλλαγών βουλευτών. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, στρατηγικής δέσμευσης και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε την κοινή κατανόηση για κάποια ζητήματα και να ενισχύσουμε επίσης τη συνεργασία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ βουλευτών από τις δύο πλευρές και χαιρόμαστε πάρα πολύ διότι τρει επιτροπές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρθαν ήδη στο Κοινοβούλιο τη Συνδικής τη διάρκεια του 2017 και εκτιμούμε πάρα πολύ την πρόσκληση που μα είχε απευθύνει ως πρέσβης για την Ινδία από τότε που ανέλαβα το αξίωμά μου τον Ιούλιο έκανα πολλέ απόπειρε και προσπάθειες και εν τέλει μίλησα με τον αρμόδιο υπουργό μα στο Νέο Δελχή πριν από μερικέ εβδομάδε, η οποία μα είπε ότι στα πλαίσια του δικού μα συστήματο η μόνιμη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων δεν προβλέπει ταξίδια στο εξωτερικό. Αυτή είναι η παράδοση που ακολουθείται στη χώρα μου. Παρ' όλα αυτά δεν πρόκειται να εγκαταλείψω την προσπάθεια, σας το υπόσχομαι. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα καταφέρω να φέρω κάποιους σημαντικούς βουλευτές από το δικό μας το κοινοβούλιο προκειμένου να έρθουν και να σας μιλήσουν εδώ πέρα. Μας έχετε κάνει την πρόσκληση αυτή, την έχετε επαναλάβει πολλές φορές, την εκτιμούμε όλους ιδιαιτέρως και θεωρώ πραγματικά ότι θα πρέπει με τον έναν άλλο τρόπο η επίσκεψη αυτή από το Κοινοβούλιο της Ινδίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει χώρα. Είναι σε εξέλιξη, αν θέλετε, η όλη δική μου προσπάθεια. Να απαντήσω καταρχάς στις ερωτήσεις του κυρίου Νταν Πρέντα. Σας ευχαριστώ πολύ για το ρόλο που έχετε διδραματίσει ως συγητής κατά την εκπόνηση του εξαιρετικού αυτού ψηφίσματος για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας να επενθυμίσω ότι ε, αναφερθήκατε σε έναν οικονομικό διάλογο υψηλού επίπεδου. Ακριβώς αυτό ζητήσαμε και εμείς, αυτό ακριβώς θέσαμε στα πλαίσια των προτεραιοτήτων, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο την πρότασή σας αυτή για τη θέσπιση ενός τέτοιου ε, οικονομικού διαλόγου υψηλού επίπεδου. Προφανώς δεν έχουμε καταλήψει την ιδέα αυτή, την επεξεργαζόμαστε ακόμη και αυτή η διάσκεψη κορυφής, όπως το είπατε κι εσείς, εμφύσισε νέα δυναμική στην στρατηγική μας σχέση για να δανειστώ και κάτι που είπε ο κύριος ε, Γιούνκερ, πραγματικά πνέει νέος άνεμος στα πανιά της, σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία. Αυτό αληθεύει όπως είπε και ένας από τους προλαλήσαντες, είναι ιδιαίτερα μακροσκελής η διακήρυξη αυτή, η δήλωση που γίνεται. Αναφερθήκατε στη δυνατότητα να έχουμε έναν οδικό χάρτη για την εξέλιξη των σχέσεών μας. Εγώ θεωρώ ότι αφού καταφέραμε μετά από μια μεγάλη περίοδο πραξίας να καταλήξουμε σε δύο συνόδους, ήταν πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε και μία δήλωση κοινή, ακόμα και μακροσκελή, προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να έχουμε έναν πιο λεπτομερή και πιο πλήρη οδικό χάρτη. Και απαντάω κατά αυτόν τον τρόπο και σε μια άλλη ερώτηση που έγινε από έναν Ευρωβουλευτή πριν από λίγο. Α προσεγγίσουμε λοιπόν την κοινή αυτή δήλωση, μολονότι είναι μακροσκελή και ιδιαίτερα λεπτομερή, ω ένα οδικό χάρτη επί του οποίου έχουν συμφωνήσει και οι δύο πλευρέ. Αναφερθήκατε επίση στην κρίση στο Μιανμάρ. η Ινδία από την πρώτη και όλα μέρα της κρίσης αυτής για τους Ροχίνγκια ζήτησε να ενημερωθεί για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση επιτόπου. Μας ανησύχησε όλους ιδιαίτερο το ζήτημα αυτό και άμεσα διοργανώσαμε την αποστολή ενός σκάφους με ανθρωπιστική βοήθεια που θα έφτανε στο Μιανμάρα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τον Μπαγκλαντές με το οποίο συνεργαζόμαστε πολύ στενά προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι Για κάθε εκτοπισμένο άτομο θα προβλέπεται ένα δέμα με τρόφιμα, με νερό, με κάποια είδη πρώτης ανάγκης και έχουμε αποστείλει τα δέματα αυτά τα οποία πήγανε προς τους αποδέκτες τους, τα άτομα αυτά τα οποία βρίσκονται στους καταβλισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόκειται για μια βοήθεια δική μας η οποία διοχετεύεται μέσω της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές, καθότι είναι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές εκείνη η οποία υποδέκτηκε τα εκτοπισμένα αυτά άτομα στην επικράτειά της. Στείλαμε λοιπόν και σκάφη και αεροσκάφη με την ανθρωπιστική αυτή βοήθεια, με τα θέματα αυτά τα οποία σας ανέφερα. Θεωρούμε ότι η ανθρωπιστική αυτή κρίση θα πρέπει να επιληθεί μέσω ενός ειλικρινούς διαλόγου και ότι θα πρέπει με οριμότητα και ιδιαίτερη προσοχή να διευθετήσουμε το ζήτημα. Θεωρούμε ότι μία μέθοδος, αν θέλετε, θα ήταν να καταφέρουμε να πετύχουμε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στην επαρχία του Ρακίν και μάλιστα συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση της Μιανμάρ προκειμένου να έχουμε ένα αναπτυξιακό πλέον ταμείο για την επαρχία του Ρακίν, καθότι θεωρούμε ότι αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στο να επιστρέψουν στην επαρχία του Ρακίν τα εκτοπισμένα αυτά άτομα τα οποία βρίσκονται εκτό Μιανμάρ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα στι 9 Σεπτεμβρίου προχωρήσαμε σε μία επίσημη δήλωση. Ο Πρωθυπουργό μα είχε πάει στο Μιανμάρ τι προηγούμενε μέρε και αμέσω μετά την εμφάνιση των γεγονότων αυτών και στη δήλωσή του αναφέρθηκε επίση τη γενικότερη ανησυχία που τρέφουν οι ηγέτε παγκοσμίω αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άσκησε πίεση στην κυβέρνηση τη Μιανμάρ να ασχοληθεί με το ζήτημα των Ροχίνγκια και να βρεθεί τελικά μια λύση βάσει της δικαιοσύνης, της ειρήνης, αξιοπρέπειας και των δημοκρατικών αξιών. Και όπως σας είπα, εμείς σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Μιανμάρ θέλουμε να συμβάλλουμε περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη της επαρχίας του Ρακίν και ο Πρωθυπουργό μας συνομίλησε μάλιστα και με την Άουν Σαν Σοουκή και άσκησε πίεση στην κυβέρνηση της Μιανμάρ, λέγοντας ουσιαστικά ότι όλος ο πλανήτης πλέον ανησυχεί για την τραγική αυτή βάναυση μετατόπιση χιλιάδων ατόμων Ροχίνγκια και θεωρήσαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να σταματήσει η βία και να αποκατασταθεί η τάξη το συντομότερο δυνατό και μάλιστα προσπαθήσαμε με προσοχή και οριμότητα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή, λέγοντας ότι θα πρέπει να προασπίσουμε στο δυνατόν περισσότερο τους εκτοπισμένους αυτούς πληθυσμούς, αναφερόμενοι βέβαια και στις δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρα. Πώς μπορούμε τώρα να επιλύσουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση την κρίση αυτή. Δεν έχει αποτανθεί κάποια επίσημη πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεργαστούμε από κοινού για την, για την κρίση των Ροχίνγκια. Πάντως, όταν οι αρμόδιες αρχές μας συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούγκερ, είχαμε θίξει και το ζήτημα αυτό στα πλαίσια της Συνόδου, ότι θα πρέπει δηλαδή να συνεργαστούμε για να επιλύσουμε το πρόβλημα με τη μειονότητα των Ροχίνγκια. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Βανόρντεν, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ θετικά, θερεντικά σας λόγια. Ως πρέσβης της Ινδίας είναι πραγματικά προνόμιο για μένα να μπορώ να συνεργάζομαι με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μπορώ πραγματικά να λαμβάνω τις δικές σας παρατηρήσεις, απόψεις, συμβουλές και προτάσεις και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που είχα την ε, δυνατότητα να σας συναντήσω όλους, μολονότι έχετε πολλές ανελημμένες υποχρεώσεις, ε, αφιερώστε τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να μου πείτε περισσότερο τι σας ενδιαφέρει σε σχέση με τις ε, σχέσεις που έχουμε Ινδία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα προσπαθήσω να προωθήσει ω βασική προτεραιότητα τη στρατηγική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ινδία. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ άλλωστε. Τόσο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η δική μου η πρεσβεία, αποτιμώντας τα αποτελέσματα τη συνόδου αυτή, θεωρήσαμε ότι ε, ανακαλύπτουμε εκ νέου ημέν τους δε. Ακόμα και ο πρόεδρο Τούσκ τον έφερε αυτό στι ε, δηλώσει που έκανε αφού του επέστρεψε από τη σύνοδο αυτή και μάλιστα είπε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να προωθήσει πολύ πιο δυναμικά την εταιρική σχέση Ινδίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά θα ήθελα και εγώ να πω ότι από τη δική μου την πλευρά θα ανταποκριθώ στην νέα αυτή δυναμική που διαφαίνεται τώρα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα κονδύλια τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει πλέον ένα γραφείο στο Νέο Δελχή και αυτό αποτελεί έμπρακτη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Ινδία. Η χρηματοδότηση των βασικών υποδομών μας είναι πάρα πολύ σημαντική και θα θέλαμε με τρόπο αποτελεσματικό να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να ευοδοθούν αυτές οι επενδύσεις. Τώρα, μας ρωτήσατε αν είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι, τι γίνεται με τις τομεακές συμφωνίες και αν όντως μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια πλήρη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Όντως υπάρχει μια έντονη πολιτική βούληση, ο δικός μας ο Πρωθυπουργό είπε ο ίδιος ότι ε, έχουμε κάνει ένα υπαρκή απολογισμό της κατάστασης και ότι θα πρέπει πλέον να προχωρήσουμε σε έμπρακτη δραστηριοποίηση. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής, ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ είπε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις αφού βέβαια πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Όταν λίγο αργότερα συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τους ρωτήσαμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό όταν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως είπε ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί εμείς ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω διαπραγματεύσεις. Οι επαρκείς λοιπόν αυτές προϋποθέσεις συζητήθηκαν στις 13 και 14 Νοεμβρίου. Είχαμε μία επίσκεψη της ε, επικεφαλής διαπραγματεύσεων από την ευρωπαϊκή πλευρά, η οποία ήρθε στην Ινδία με την ε, διαπραγματική ομάδα και συζητήσαμε όλες τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει χώρα στην Ινδία και που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Από το 2013 και μετά, ξέρετε ότι το 2013 ήταν ο τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων, προσπαθήσαμε να δούμε τι έχει γίνει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων, στο ζήτημα των περιορισμών που υπήρχαν όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, τι δημόσιε συμβάσει και αποφασίσαμε να προωθήσουμε τα ζητήματα αυτά στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου πλέον χρονοδιαγράμματος. Ήταν πολύ σημαντικό το να καταφέραμε και οι δύο πλευρές να φερθούμε στα ζητήματα αυτά. Είδαμε ποιε ήταν οι απαιτήσει και προσδοκίες από κάθε πλευρά. Η ευρωπαϊκή πλευρά ήταν πιο συγκρατημένη στη φιλοδοξία της. Εμείς από τη δική μας την πλευρά προσπαθήσαμε να θέσουμε τους δικούς μας φιλοδοξού στόχους και αποφασίστηκε εν τέλει ότι μέχρι τα τέλη του ε, τέταρτου τριμήνου του 2018 θα πρέπει να συναντηθούμε εκ νέου και να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτές οι συναντήσεις, οι γύροι διαπραγματεύσεων τελικά, κατέληξαν σε μία ημερομηνία για την επόμενη μας συνεδρίαση, κατέληξαν σε συγκεκριμένη ανακοίνωση για τους τομείς επί των οποίων θα συνεργαστούμε και προσέδωσαν μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες αυτές τις συζητήσεις και έπειτα είχαμε και κάποιες επιμέρους ομάδες εργασίας για επιμέρους ζητήματα συζητήσαμε πάλι εκ νέου για τομιακά πλέον ζητήματα στις 14 Νοεμβρίου και στα πλαίσια των ομάδων αυτών εργασίας προσπαθήσαμε να επιλύσουμε προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει στο παρελθόν όσον αφορά την τομιακή μας αυτή συνεργασία. Πάλι επιδείξαμε επικοδομητικό και θετικό πνεύμα προκειμένου να απομπλοκαριστεί η κατάσταση. Εγώ λοιπόν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη, έχοντα δει πώ εξελίχθηκαν οι τελευταίε αυτέ συζητήσει 13, 13 και 14 Νοεμβρίου και συμφωνώ με εσά ότι έχουμε καταπληκτικές ευκαιρίες στο μέλλον, ιδίως στα πλαίσια της τωρινής συγκυρίας και επικεντρωνόμαστε και εμείς πάρα πολύ στην σχέση που θα έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Τάνοκ τώρα σας ευχαριστώ και εσάς. γιατί όντως ξεκινήσατε εσείς τον όλο διάλογο Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη σύσταση τη ομάδα των φίλων τη Ινδία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι είχαμε κάτι τέτοιο και συνέβαλε πάρα πολύ στο να ενισχυθούν οι σχέσεις ανάμεσα στα δύο κοινοβούλια και ε, εγώ ανέκαθεν θεωρούσα ότι ήμασταν φίλοι και στις 25 Οκτωβρίου είχα τη δυνατότητα να σας μιλήσω στο Στρασβούργο και είχα τη δυνατότητα να δω επίση ποιοι είναι οι βασικοί τομεί προτεραιότητα που σα ενδιαφέρουν. Αναφερθήκατε στο Mode 4, αναφερθήκατε επίση στο Brexit και είπατε επίση ότι ε, θα μπορούσαμε να κινηθούμε πιο γρήγορα σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Όντω, το Mode 4 είναι ένα σημείο επί το οποίο θα πρέπει να συνεχιστούν περισσότερο οι συζητήσεις μας, σημείο το οποίο θα πρέπει να επιλύσουμε και θα πρέπει τελικά να καταλήξουμε σε μία λύση επωφελή και για τις δύο πλευρές. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο σε αυτό το ζήτημα. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούμε να προδικάσουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μετά το Brexit. Παρακολουθούμε προσεκτικά πώς θα διαμορφωθούν οι όροι αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας πολύ σημαντικός παραδοσιακός εταίρος της Ινδίας, μακρόχρονη η σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος. Θα εξετάσουμε λοιπόν κάθε μία από τις σχέσεις αυτές προσεκτικά και ξεχωριστά και είμαστε πεπισμένοι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσουν να έχουν κατά νου και στο μέλλον πόσο σημαντικό είναι για μας, για τους Ινδούς, να μπορούμε να έχουμε μια πιο έντονη κινητικότητα των επαγγελματιών μας. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της οικονομικής μας συνεργασίας. Να αναφερθώ τώρα και στις παρατηρήσεις του κυρίου Μπούχνερ Πραγματικά μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπάρχουν μεταπτυχιακοί φοιτητέ από την Ινδία στη Γερμανία. Εγώ νόμιζα ότι όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα παντού στον κόσμο είχαν τουλάχιστον 10 και παραπάνω Ινδούς μεταπτυχιακούς φοιτητέ. Θα ασχοληθώ λοιπόν προσωπικά με το ζήτημα αυτό, θα έρθω εκ νέου σε επαφή μαζί σας και θα έρθω σε επαφή επίσης με το αρμόδιο Υπουργείο στην ε, Ινδία, καθώς επίσης και με τα πανεπιστήμια μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να έχουμε ανταλλαγές φοιτητών σε κάθε περίπτωση. Εμείς καλωσορίζουμε στην Ινδία πολλούς ξένους φοιτητές και ο Πρωθυπουργό μας έχει ε, αποτείνει έκκληση προς τους φοιτητές διαφόρων χωρών, προκειμένου να μπορούμε τελικά σε όλα τα επίπεδα να έχουμε παρουσία ξένων φοιτητών. Ξέρετε ότι υπάρχουν διάφοροι τομεί, όπω η ιατρική για παράδειγμα, όπου θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να, έχουμε, έχουμε περισσότερου φοιτητέ από το εξωτερικό. Μπορούμε κι εμεί όμω από τη δική μα την πλευρά να συμβάλλουμε πάρα πολύ στον τομέα τη επιστήμη, τη τεχνολογία, στον τομέα τη μηχανική, στον τομέα τη καινοτομία. Να συμβάλλουμε πάρα πολύ στη δημιουργία νεοφιών επιχειρήσεων. Και προφανώ θα θέλαμε κι εμείς να καλωσορίσουμε στην Ινδία ταλαντούχου νέου από όλε τι περιοχέ του κόσμου. Θα ήθελα λοιπόν να συνεργαστώ περαιτέρω μαζί σας στους τομείς αυτούς που θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ανταλλαγή φοιτητών και να έχουμε περισσότερους Ινδούς φοιτητούς, φοιτητές με συγχωρείτε και στη Γερμανία. Δεν ξέρω να απάντησα σε όλα τα ερωτήματα και σε όλες τις παρατηρήσεις κλιματικές αλλαγές. Ναι, ναι. Η κοινή μας δήλωση έχει τρία εδάφια τρεις παραγράφους για την κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να το σημειώσετε αυτό. Μας ανησύχησε ιδιαίτερα η μόλυνση στην πρωτεύουσα από την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου και υπάρχουν και κλιματικοί λόγοι από ό,τι φαίνεται πλέον. Κάποιοι συγκεκριμένοι άνεμοι που πνέουν από τις ερήμους Αλλά βεβαίως είναι επίγουσα ανάγκη να ρυθμίσουμε, να, να λάβουμε μέτρα για τη μόλυνση αυτή. Είμαστε μέλος και της Solar Alliance. Η αιωλική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές είναι υψηλής προτεραιότητας για εμάς. Μπορώ να σας δώσω την ερχόμενη εβδομάδα πολύ περισσότερε λεπτομέρειε για το τι κάνουμε στα πλαίσια κλιματική αλλαγή. αλλά έχουμε φιλόδοξου στόχου. μπορώ να σα βεβαιώσω, έχουμε εθνικά προγράμματα, στόχου. και οπωσδήποτε είναι μια περιοχή υψηλωτά τη προτεραιότητα για εμά. Ευχαριστούμε την κυρία Πρέσβη. Ε, με ενημερώνουν ότι οι συνάδελφοι από τα Δυτικά Αλβάνια περιμένουν έξω από την αίθουσα. Θα πρέπει να μην τους καθυστερήσουμε πολύ περισσότερο. Αν θέλετε σε ένα λεπτό να συνοψίσετε. Ναι, οπωσδήποτε, Πρόεδρε, θέλω να μακρηγορήσω και να σας καθυστερήσω. Και βεβαίως η κυρία Πρέσβης τα είπε όλα ή σχεδόν όλα. Δύο κουβέντες θα προσθέσω και εγώ και ίσως τα γαλλικά αν μου επιτρέπετε για τα στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής έχουμε μια κοινή δήλωση πολύ φιλόδοξη και πληρέστατη. Και συμφωνώ απολύτως με την κυρία Πρέσβη επί του ότι η ευρύτητα του κειμένου είναι και αυτή μια ένδειξη της βαρύτητος της σχέσης. Και θα δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ένα φιλοπορίας ε, για τη συνέχεια θα μπορούσαμε ίσως να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι για τα θέματα της Ουκρανίας, των Ροχίνγκια. Νομίζω όμως ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά ενεργή στο θέμα αυτό και με την πρόσθετη επίσκεψη της ε, είπα εκπροσώπου και μαζί με την ε, Σύνοδο των Υπουργών και τη συνάντησή τους ε, με τις χώρες ΑΣΕΜ Νομίζω ότι συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες της άλλης πλευράς και παρότι μπορεί να μην έχουμε συγκεκριμένα έργα, προγράμματα συνεργασίας ε, και εμείς συνδιοργανώσαμε στη Γενέβη την ε, διάσκεψη των δωρητών, επομένως η δέσμευσή μας είναι σαφής. Για την φιλοδοξία την εμπορική δεν έχω παρά να αντιχίσω τα όσα είπε η πρέσβης, και απλώς θα πρέπει να καθορίσουμε ένα κοινό επίπεδο φιλοδοξίας προκειμένου να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα αυτών. Για την κλιματική αλλαγή και προσπαθώ να διατρέξω διάφορα παραδείγματα όπου έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία μας υπάρχει μια σειρά από περιοχές που προσπαθούμε να προχωρήσουμε. Είμαστε ήδη πολύ ενεργητικοί στη συνεργασία αυτή. Ε, ανέφερα τη Διεθνή ε, Συμμαχία για τον Ήλιο και η Ινδία ενδιαφέρεται να προχωρήσει στα θέματα της ηλιακής ενέργειας. Η συνεργασία με τις τοπικές αρχές, η Σύνοδος των Δημάρχων, το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι και αυτό ένα παράδειγμα στα πλαίσια του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί βέλτιστες πρακτικές και συνεργασία. Έχουμε διάφορες πιλωτικές επισκέψεις, ο Επίτροπος Βέλα, Άγιες ε, ε, προτίθεται να επισκεφθούν την Ινδία στο άμεσο μέλλον. Θα σταματήσω εδώ για να μην καθυστερήσω αλλά νομίζω ότι στα πλαίσια του Εράσμους η Ινδία είναι ο καλύτερος μας πελάτης στο Εράσμους Plus, αν μπορώ να το πω έτσι. Έχουμε πολλούς Ινδούς φοιτητέ και, θα... και ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε. Ευχαριστούμε την κυρία Ντελάτρε, ευχαριστούμε την κυρία Πρέσβη. Είχαμε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Ενημερωθήκαμε όλοι για το καθεστώς των συζητήσεων των σχέσεων Ινδίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Χωρίς άλλη καθυστέρηση πάω απευθεία στο επόμενο σημείο αν θέλετε να εισέλθουν οι προσκεκλημένοι μας.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

Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, με μία μικρή καθυστέρηση περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το υπαριθμό 10, το, η διάμεση αναθεώρηση του προενταξιακού μηχανισμού αντιστοίχηση χρηματοδότησης με πολιτικές προτεραιότητες. Σας καλωσορίζω και καλωσορίζω και τους προσκεκλημένους μας από τα Δυτικά Βαλκάνια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος ε, που σας δεχόμαστε στην σημερινή μας συνεδρίαση. Για τους συναδέλφους από τα Δυτικά Βαλκάνια, μια σημαντική πληροφορία για τις γλώσσες η μακεδονική ακούγεται στο κανάλι 17, η σερβική στο κανάλι 10, η αλβανική στο κανάλι 27, η βοσνιακή στο κανάλι 10, όπως και η μαυροβουνιακή γλώσσα. Πρόκειται λοιπόν για μια συζήτηση για το μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας για τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο μας απασχολεί συχνά στην Επιτροπή μας. Και βεβαίως το απόγευμα θα συναντηθούμε με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, την ευρύτερη, για το ευρύτερο θέμα της ολοκλήρωσης. Σήμερα το πρωί λοιπόν θα συζητήσουμε την οικονομική πτυχή. Καλωσορίζω και τους σημερινούς ομιλητές, ε, την κυρία Μαρίτια Σχάκε πρώτα απ' όλα από την Ολλανδία και την Άλντε, τους φιλελεύθερους, ε, που καλύπτει τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα. Κατόπιν ε, την κυρία Λουίς Καλαβέρα, διευθύντρια των Δυτικών Βαλκανίων το εκτελεστικό κομμάτι της εξωτερικής υπηρεσίας και τέλος τον κύριο Ρίφερε, ερευνητή ευρωπαϊκών πολιτικών. Σήμερα λοιπόν στόχο έχουμε να δούμε τις προοπτικές για το πώς θα αυξηθεί η αξία της χρηματοδότησης της περιοταξιακής βοήθειας. Θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι θέτουμε πολιτικές προτεραιότητες, παρακολουθούμε την εφαρμογή και τα αποτελέσματα. Και βεβαίω για να βλέπουν οι πολίτες αυτά αποτελέσματα πρέπει να ενημερώνουμε τους τελικούς δωρητές οι οποίοι είναι οι πολίτες μας για το από πού προέρχεται η χρηματοδότηση. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να δούμε αν είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί, αν βοηθάμε τα Δυτικά Βαλκάνια να έρθουν πιο κοντά στην Ένωση και τι και πώ πρέπει να βελτιωθεί. Και βέβαια θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διοικητική συνεργασία για να ενισχυθεί ε, και η ικανότητα της διοίκησης να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα και βεβαίως να δημιουργηθεί ένας βιώσιμος ενάρετος κύκλος και τι μαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε από το δεύτερο μισό της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου και μετά το 2020 βεβαίως. Σας καλωσορίζω λοιπόν να πω ότι έχουμε δώσει κάρτες στους συναδέλφους από τα Δυτικά Βαλκάνια για να μιλήσετε. Δώστε τις λοιπόν στην γραμματεία. Υπάρχει άλλη μια ανακοίνωση. Ε, πείτε τα εσείς, δεν μπορώ άλλο. σερβικά, βοσνιακά και μαυροβουνιακά βγαίνουν από το 26 παρά το ότι είναι διαφορετικές γλώσσες. Τον λόγο λοιπόν δίνω πρώτα στην κυρία Μαρίτια Σχάκη. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας καλωσορίσω και εγώ. Χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα τεχνικό και επίκαιρο θέμα, τα προενταξιακά κονδύλια για να δούμε πώς ακριβώς ε, δαπανώνται και αν υπάρχει σωστή υποκτία. Βεβαίω συμμετέχω στην ομάδα εργασία για τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα και συνομιλώ με την Κομισιόν, με τους αποδέκτες, με την κοινωνία των πολιτών. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτή η γενική εικόνα του ποιο ε, συμμετέχει σε αυτά τα ταμεία θα μας ε, δώσει μια εικόνα του γενικότερου πλαισίου. Επίσης, να αναφερθώ και εγώ σε αυτό το οποίο είπε ο Ντέιβιντ, ότι κάθε ευρώ που ξοδεύεται πλέον ελέγχεται πάρα πολύ αυστηρά, μιλάμε για δημόσιο χρήμα και πρέπει άρα να λέμε σαφώς το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Από τη μία λοιπόν μπορεί να πει κανείς ότι η προενταξιακή βοήθεια και το σχετικό μέσο έχει έναν ξεκάθαρο στόχο, το οποίο, ο οποίος είναι ακριβώ ε, να βοηθηθούν οι χώρες για να ενταχθούν. Αλλά ε, το μέτρο της επιτυχίας δεν μπορεί να είναι μόνο η ένταξη αυτών των χωρών. Υπάρχουν πολλά στάδια καθοδών προς την ένταξη, τα οποία πρέπει να τα δούμε βήμα-βήμα και χώρα-χώρα, γιατί στην πραγματικότητα για τις περισσότερες ε, από αυτές τις ε, χώρες η ένταξη ακόμα απέχει πολύ και μάλιστα είναι εκτός του πλαισίου του τρέχοντος ε, χρηματοδοτικού πλαισίου. Οπότε ο προϋπολογισμός αυτός υπό τον μηχανισμό πενταξιακής βοηθείας αλλά και άλλα πλαίσια έχουν βραχυπρόθεσμους στόχους και συγκεκριμένα παραδοτέα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο για να μπορούμε να μετρήσουμε την επιτυχία και να δούμε τα σημεία εφαρμογής αυτών των στόχων. Αν έχουμε έναν καλύτερο στόχο θα μας επιτρέψει να έχουμε και ευελιξία, να προσαρμοζόμαστε δηλαδή στις συνθήκες που αλλάζουν στις ε, χώρες, αλλά και να δούμε τα ζητήματα αυτά με τρόπο πιο συνεπή. Βεβαίω, η υπόσχεση more for more πάντα υπάρχει. Δηλαδή μια χώρα που τα πάει καλά ανταμείβεται, ενώ αν υπάρχει οπισθοχώρηση, ίσως υπάρξει προσωρινή αναστολή των κονδυλίων, τα οποία θα διοχετευτούν αλλού, παραδείγματος χάρη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αντί για κρατικούς φορείς. Ο τρέχον κανονισμός μάλιστα ανταμείβει την, απόδοση για να υπάρχει κάποιο κίνητρο. Ταυτόχρονα έχει γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί ένας τρόπος να μετρηθεί η πρόοδος, βλέποντας κάποια μέτρα και δείκτες απόδοσης. Είναι μια εξέλιξη που θεωρώ ότι πρέπει να συνεχιστεί και προς τα εκεί πηγαίνει το Κοινοβούλιο. Και αν δεν κάνω λάθος, θα έχουμε μια αναθεώρηση των ε, δικτών απόδοσης πριν το τέλος του έτους. Λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν για τα μετρήσιμα στοιχεία. Είπα ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσουμε ακριβώς την ε, επιτυχία στην επίτευξη των στόχων, αλλά και να υπάρχει και μια υποπτία τη εκταμείευση των κονδυλίων. Αυτό είναι λογικό από την πλευρά της λογοδοσίας, ειδικά αν δούμε το σύνολο των μέσων αυτών, μιλάμε για δισεκατομμύρια το χρόνο που ξοδεύονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από πολλέ περιπτώσει που άκουσα από του ενδιαφερόμενους, αλλά και εξωτερικέ εκθέσεις αξιολόγησης, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα για να έχουμε μια ενιαία εποπτεία και ένα σύστημα αξιολόγησης και νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε την πρακτική σκοπιά των χωρών που λαμβάνουν τη χρηματοδότηση. Ε, το τρέχον σύστημα φαίνεται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τακτικές αξιολογήσεις του εάν ξοδεύονται αποτελεσματικά τα κονδύλια. Ε, Κομισιόν βεβαίως κάνει εκθέσεις προόδου αναχώρα και πολιτικές εκθέσεις, είναι δύσκολο να συνδέσουμε την πρόοδο ή την οπισθοχώρηση με την χρηματοδότηση που πηγαίνει στο μέσο προενταξιακής βοήθειας. Οπότε, ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης νομίζω ότι είναι μια αναγκαία προτεραιότητα στο μέλλον. Μετά. Λίγα λόγια για την θεσμοποίηση της ε, κοινοτικής πολιτικής. Ο γενικός στόχος της πενταξιακής βοήθειας είναι σαφής, αλλά οι στόχοι των μεμονωμένων εγγράφων είναι σχετικά ασαφείς. Ταυτόχρονα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν δίνουμε τα κονδύλια στους σωστούς κλάδους. Παραδείγματο χάρη θα πρέπει να στηρίξουμε την γεωργία ή να εστιάσουμε σε μακροπρόθεσμα έργα υποδομών για να απτυχθούν και οι χώρες αυτές αλλά και να εντεχθούν περιφερειακά. Νομίζω ότι στα Δυτικά Βαλκάνια εδώ είχαμε μια χαμένη ευκαιρία να εστιάσουμε δηλαδή περισσότερο σε μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική ε, των κονδυλίων που ξοδεύουμε. Και θα ήθελα εδώ πέρα να ακούσω την άποψή σας και για τα έργα υποδομών. Βεβαίω για εμάς ε, εδώ στην Ευρώπη αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να βοηθήσουμε προς την καλύτερη διακυβέρνηση, βελτίωση της δικαιοσύνης και τέτοια πράγματα. Τώρα νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε μια τάση, μια συμφέρουσας αλλαγή ε, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Παραδείγματο χάρη, ανταποκρινόμενοι στις ανησυχητικές εξελίξεις στην γειτονιά μας, η παγκόσμια στρατηγική μας έκανε μια αλλαγή και πήγε προς αυτό το οποίο λέμε αρχές με ρεαλισμό και βέβαια λαμβάνουμε υπόψη και τα εσωτερικά συμφέροντα της Ένωσης και αυτό συμβαίνει συνεχώς στην πράξη. Εστιάζουμε περισσότερο σε ζητήματα όπως η ασφάλεια, η διαχείριση της μετανάστευσης και φεύγουμε από την εξωτερική πολιτική, την ρυθμιστική που βασίζεται στις αρχές της Ένωσης και νομίζω ότι η παρατήρηση αυτή φάνηκε και στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών που περιγράφουν επιλέξει ότι τα τελευταία χρόνια η εστίαση είναι περισσότερο στις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι των χωρών εταίρων. Θέλω λοιπόν ότι οι ανάγκες ε, των πρωτεξιακών χωρών και των κρατών μελών είναι αλληλένδετες. Αν δούμε τα Δυτικά Βαλκάνια, αν δεν πάνε καλά αυτές οι χώρες, σαφώς επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν μπορούμε να απομονώσουμε τα εσωτερικά συμφέροντα της Ένωσης από την ευημερία των ανθρώπων και τις δημοκρατικές εξελίξεις στις χώρες αυτές. Και βεβαίως ε, εκεί πέρα έχουν σύνδεση και οι πολιτικές προτεραιότητες. Επίσης ε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην ταυτίσουμε τις χώρες ε, σε σχέση με το τι ζητάνε οι κυβερνήσεις, αλλά να θέσουμε τον λαό τους ε, σε πρώτη μοίρα. Θα αναφερθώ τώρα σύντομα στην κατάσταση που βλέπουμε στην Τουρκία, γιατί έχει γίνει το κύριο θέμα ε, που απασχολεί το Κοινοβούλιο και ίσως υπάρχουν και κάποια μαθήματα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Ερντογάν η χώρα κατευθύνεται προς μια αυταρχική ε, κατεύθυνση. Συλλαμβάνονται ηγέτες αντιπολίτευσης, ε, δημοσιογράφοι, χωρίς κατηγορίες, αλλά βλέπουμε προσπάθειες ε, για να υπάρξει συγκεντρωτισμό στην εξουσία μέσω της αναθεώρησης του συντάγματος, που θα σημαίνει ότι η Τουρκία δεν πληρεί πλέον τα κριτήρια της Κοπεχάγης. Οπότε το ερώτημα του εάν η πενταξιακή βοήθεια πρέπει να συνεχιστεί έχει ακουστεί τουλάχιστον εδώ μέσα και ακούγεται όλο και πιο δυνατά. Ταυτόχρονα υπάρχει σαφής ανάγκη να βοηθήσουμε τον κόσμο στην Τουρκία, να ενισχυθεί η ελευθερία των ΜΜΕ και οι λοιποί πυλώνες. Οπότε αυτό το οποίο είναι σημαντικό να σημειώσουμε είναι ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή το θεσμικό πλαίσιο για το προενταξιακό μέσο είναι πολύ ακαμπτό και καθιστά δύσκολο το να ανακατευθύνουμε αλλού αυτά τα κονδύλια παρά το ότι υπάρχει η πολιτική βούληση. Δεύτερον, υπό το πρίσμα της λεγόμενης συμφωνίας ή δήλωσης για την Τουρκία βλέπουμε ότι τα λεφτά από διάφορα εξωτερικά κονδύλια έχουν ανακατευθυνθεί για την διαχείριση της μετανάστευσης και αυτό δείχνει ότι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο αρκεί να συμφωνήσουν οι αρμόδιοι φορείς όχι μόνο μόνο για την μετανάστευση, αλλά να δούμε και τον αντίκτυπο στην περιοχή και τους μακροπρόθεσμους στόχους. Επίσης, να σημειώσω το Κοινοβούλιο δεν ερωτήθη για την σύμφωνη γνώμη του για την δήλωση με την Τουρκία, παραδείγματος χάνει, για τη μετανάστευση. Θα καταλήξω με λίγα λόγια για τη μασοπρόθεσμη αναθεώρηση. Ήθελα να τονίσω την περίπτωση της ε, Τουρκίας για να έχουμε μια αίσθηση της δυναμικής ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως ένα παράδειγμα όπου βλέπουμε ότι είναι δυνατή ανακατεύθυνση των κοντιλίων αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση αλλά υπάρχει κάποιο χάσμα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Ελπίζω ότι με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την αξιολόγηση της δυναμικής με τις χώρες της γειτονίας θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και το τι πρέπει να κάνουμε στο θεσμικό πλαίσιο, στα μέτρα σύγκρισης, ε, στην εποπτεία, οπότε αναμένω τη σημερινή συζήτηση που νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση που θα παρουσιάσει η Κομισιόν τον Σεπτέμβριο. Ελπίζω λοιπόν να συνεχιστεί η χρηματοδότηση για τα επόμενα δύο έτη και να μπορούμε να μιλάμε και για πέρα από αυτή την περίοδο μετά το 2020. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και αναμένω τη σημερινή συζήτηση. Thank you. Ευχαριστούμε την κυρία Σχάκε για τα εισογικά της σχόλια. Πάμε τώρα στον κύριο, στην κυρία Ρουίθ Καλαβέρα που εκπροσωπεί εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Μακάλιστερ, ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση αυτή. Εχθές είχα ένα δείπνο με τους εκπροσώπους της Βοσνίας και αλλά θα ήθελα να καλωσορίσω με την ευκαιρία αυτή τους εκπροσώπους όλων των χωρών της περιοχής. Βλέπω και κάποια γνώριμα πρόσωπα, τον πρώην Υπουργό Χότσι, αν ακούσαμε καλά το όνομα, είναι νομίζω απολύτως επίκαιρη η στιγμή τη συζήτηση του προενταξιακού μέσου, γιατί αυτή τη στιγμή σημειώνουμε, καταγράφουμε τα όσα έχουμε επιτύχει τα προηγούμενα χρόνια και προετοιμάζουμε και την ενδιάμεση, την μεσοπρόθεσμη μάλλον επανεξέταση. Έχουμε εξωτερική αξιολόγηση όλων των μέσων από ανεξάρτητους εξωτερικούς δηλαδή αξιολογητές και τώρα πλέον η Επιτροπή θα εξετάσει όλα αυτά τα πορίσματα, όλες αυτές τις μελέτες προκειμένου να προχωρήσει σε μια δική της εκτίμηση αντικτύπου. Θα υποβληθεί ένα έγγραφο τον Δεκέμβριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα είναι η βάση της συζήτησης που θα πλαισιώσει το στρατηγικό μας διάλογο από νωρίς του χρόνου. Τα υπόλοιπα χρόνια δηλαδή που έχουμε υπό τις παρούσες προοπτικές. Ο IPA κανονισμός συμπεριλαμβάνει 7 δισεκατομμύρια συνολικά προενταξιακής βοήθειας και αυτά αφορούν στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε η κυρία Σχάκη, να ε, εξασφαλίσουμε ότι τα μέσα αυτά θα προετοιμάσουν το έδαφος και θα προσελκύσουν επενδύσεις. Όλοι οι πληθυσμοί της περιοχής, όλα τα κράτη αυτά έχουν αγκαλιάσει αυτό το μέσο και έχουν την απαραίτητη φιλοδοξία. Όμως χρειάζεται ευθύνη από την κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση στις χώρες αυτές. Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι κρίσιμος ώστε να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες. Προς μια ενταξιακή οδό και επομένως πρέπει να μας βοηθήσετε και εσείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να εξηγουγήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αιρεσιμότητα και τις υπόλοιπες συνθήκες που συνδέονται με όλη αυτή τη χρηματοδότηση στις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις και χώρες. Τώρα, το πιο σημαντικό της εξωτερικής αυτής αξιολόγησης είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια θετικά συμπεράσματα τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Καταρχάς, ότι υπάρχει στενός σχετισμός της υλοποίησης του IPA μεταξύ των φιλοδοξιών μας και των προγραμμάτων βοήθειας. και υπάρχει και σχετισμό με τον προκάτοχο στι προηγούμενε δημοσιονομικέ προοπτικές. Έχουμε εστιαστεί στις διαθετικές αλλαγές για να βοηθήσουν και να προετοιμάσουν τι χώρες αυτές για ένταξη. Επομένως, εστιαζόμαστε στις περιοχές προτεραιότητας. Δηλαδή, στην υποστήριξη και θεμελίωση της δημοκρατίας, της μεταρρύθμισης ε, της δημόσιας διοίκησης, του κρατου δικαίου, της προστασίας των μελιωδών δικαιωμάτων, της οικονομικής ανταγωνιστικότητος και βεβαίως του να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες αυτές δεν θα προχωρούν μόνο διμερός στη σχέση τους μαζί μας, αλλά θα συνεργάζονται και περιφερειακά μεταξύ τους. Γιατί όσο καλύτερη περιφερειακή συνεργασία έχουν οι χώρες, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η όθηση προς τα εμπρός προς την κατεύθυνση της εντάξεως. Χρησιμοποίησαμε επίσης τον IPA 2 ώστε να είναι ευέλικτος και να προσαρμόζεται προς έκτακτες ανάγκες. Είχαμε πλημμύρες στη Βοσνία και καταφέραμε να κάνουμε ανακατανομή, αναπίστωση αν θέλετε των κονδυλίων βοήθειας που για να αντιμετωπιστούν οι ζημιές και οι καταστροφές τέτοιων φαινομένων. Και ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που είχαν πληγεί σε μεγαλύτερο βαθμό και από την εισρωή της μετανάστευσης. Άλλη μια πτυχή που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι η αξιολόγηση έχει σημειώσει ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο IPA καθιστά τη μόχλευσή μας πιο έντονη. ώστε να έχουμε καλύτερη προστιθέμενη αξία στο έδαφος. Ο ΑΕΠΑΗ μας έχει βοηθήσει λοιπόν στην οικονομική μας μόχλευση και στην καλύτερη υλοποίηση των χρηματοπιστωτικών ε, μέσων που ενεργοποιούμε στην περιοχή. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις συνέργειες με άλλα μέσα, όπου θα έχουμε καλύτερη συνέπεια πολιτικής ε, για την ανάπτυξη. και για μέσα τα οποία αφορούν μάλιστα στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας και των, της προστασίας των δικαιωμάτων, αυτά μπορούμε να τα δούμε σε μεγαλύτερο βάθος. Τα μέσα που έχουν σχέση με τις πολιτικές φιλοδοξίες και των χωρών και της περιοχής και, των Ευρω... και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται δηλαδή για μέσα που θα σας βοηθήσουν να γίνετε εσείς οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μελλοντικά μέλη. Δηλαδή θα σας προετοιμάσουν για να καλύψετε το έδαφος που σας χωρίζει από τη στιγμή κατά την οποία θα είστε έτοιμοι για εισδοχή. Και βεβαίως ο στόχος της ένταξης είναι ένας θα έλεγα κοινός στόχος για όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Πρέπει δηλαδή να ξεπεράσει κανείς τα στενά κομματικά συμφέροντα προκειμένου να επιτύχει το στόχο αυτό. Πρέπει λοιπόν, είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζετε τι κάνουμε με το πρόγραμμα IPA, ότι υποστηρίζετε την κατεύθυνση της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις των χωρών σας. Και το τελευταίο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι Πρέπει να δούμε τις επιδόσεις και σε τομεακό επίπεδο. Γιατί εδώ προσπαθούμε να επιτύχουμε την μεταμόρφωση, αν θέλετε, των κοινωνιών. Και στηριζόμαστε, βασιζόμαστε και στην βοήθειά σας από πλευράς εθνικών κοινοβουλίων για να εξασφαλίσουμε ότι η υλοποίηση, η εφαρμογή των προγραμμάτων στο έδαφος των χωρών σας θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις, αλλαγές στη ζωή των πολιτών. Και νομίζω από κοινού θα πρέπει να επιτύχουμε μια υψηλότερη επιφάνεια της χρήσης, της χρησιμοποίησης των ευρωαϊκών κονδυλίων. Γιατί κατά κεφαλήν είσαστε ίσως στην πρώτη θέση της βοήθειας που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές που επιχειρούμε είναι δύσκολες, το γνωρίζουμε, αλλά δεν είστε μόνοι σας. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή η χρηματοδότηση να είναι εμφανής στους πολίτες των χωρών σας και να αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δήλωσή σας. Ας περάσουμε τώρα στον τρίτο μιλητή μας, τον κύριο Φουερέ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί φίλοι. Καταρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι τα προενταξιακά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν πολύ σημαντική επένδυση για το μέλλον τόσο των χωρών εκείνων που θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο όμως και για το μέλλον της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κονδύλια αυτά έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους δικαιούχους να προχωρήσουν στις κατάλληλες οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις και να ανταποκριθούν βέβαια στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να δώσουν στους πολίτες βελτιωμένες οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες και θα πρέπει να επιτρέψουν την ανάπτυξη προτύπων που να αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία ισχύουν και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου όμως να ανταποκριθούμε στο ερώτημα το οποίο θέσατε για το πάνελ μας, και θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα αυτά που είπε ο πρώτο ομιλητή για την πολιτική διάσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώ έχει γενικότερη πολιτική κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια αυτή τη στιγμή. Όπω είπα και σε μια άλλη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου σα χθε, η περιοχή αυτή έχει οπισθοδρομήσει δραματικά. Έχει διολυστήσει σε κάθε τομέα όσον αφορά για παράδειγμα ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσμικών οργάτων, διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα. Αρκεί να θυμηθούμε την δήλωση που είχαμε στην προηγούμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική διεύρυνση για το 2016 και παραθέτω εδώ πέρα τι λεγόταν στη δήλωση αυτή, ότι η περιοχή αυτή δείχνει ξεκάθαρα συμπτώματα και πολλούς βαθμούς άλωσης του κράτους. Και βλέπουμε λοιπόν ότι οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα, ότι ήδη από το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει κάποιες θεμελιώδεις προτεραιότητες στον πυρήνα της διαδικασίας προσχώρησης. Είχαν αφαιρθεί σε ζητήματα κράτος δικαίου συγκεκριμένα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα που έχει να κάνει με τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων αλλά και άλλο, άλλες μορφές παράνομου εμπορίου συμβάλλουν όλο και περισσότερο στην αποσταθεροποίηση της περιοχής. Οι δραστηριότητες αυτές δυστυχώς βλέπουμε ότι πολλές φορές προστατεύονται από κρατικούς και πολιτικούς θεσμούς. Ορισμένοι βέβαια θα λέγαν ότι παρά την απογοητευτική αυτή ανησυχητική εικόνα, το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την εξαρτησία του δικαστικού συστήματος ή για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι είναι το πλαίσιο αυτό αρκετά υγιές και σταθερό. Αλλά αυτό απέχει πάρα πολύ από το τι συμβαίνει τελικά στην πράξη, αποτελεί μια απατηλή εικόνα της πραγματικότητας. Αυτό φαίνεται άλλωστε και στις εκθέσεις προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου λέγεται ξεκάθαρα ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι επαρκής και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη πόρων αλλά και την έλλειψη πολιτικής βούλησης. Ακόμα και θεσμικά όργανα τα οποία δημιουργήθηκαν από επιμέρους νομοθεσίες για να επιβλέπουν τις μεταρρυθμίσεις αυτές δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν και αυτό γιατί η ίδια η κυβέρνηση σε πολλές από τις χώρες Δυτικών Βαλκανίων δεν προβλέπει να δοθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι και πρέπει να υποθεί βέβαια ότι όλες αυτές οι εξελίξεις λαμβάνουν χώρα σε μια εποχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο μόνος παράγοντας στην περιφέρεια. Χθε έγινε μία αναφορά στην επιθετική εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Από την άλλη έχουμε όμως και την Τουρκία, η οποία προσπαθεί να ανακτήσει όλο και περισσότερη επιρροή στην περιοχή αυτή μέσω όλο και περισσότερων επενδύσεων. Αλλά χρησιμοποιεί επίσης και διάφορες πολιτισμικές συγγένειε, καθώς επίσης και την αυταρχική προσέγγιση που έχει όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις. Η Κίνα επίσης προωθεί όλο και περισσότερες επενδύσεις στα πλαίσια της πολιτικής «Μία ζώνη, ένας δρόμος» που ήδη ξεκίνησε από το 2013. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι οι επενδύσει αυτέ από τι χώρε αυτέ δεν λειτουργούν απαραίτητα υπέρ των χωρών αποδεκτών, δηλαδή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου κάθε φορά που Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζουμε για την κατανομή κονδυλίων στα πλαίσια του μηχανισμού προταξιακή βοήθεια. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε κάθε φορά ότι τα ζητήματα που άπτονται του κράτου δικαίου θα τίθενται πραγματικά στον ε, πυρήνα τη όλη διαδικασία. Αν αντλήσουμε διδάγματα από τον πρώτο μηχανισμό προταξιακή βοήθεια 2007, 2007 2013 που ανέφερε η προηγούμενη, η προηγούμενη ομιλήτρια και αν δούμε επίσης ε, και τους νέους στόχους που τίθενται από τον δεύτερο μηχανισμό προταξιακής βοήθειας, μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά βελτιώνονται οι επιδόσεις. Έχουμε πλέον ε, έγγραφα στρατηγικής αναχώρα που προβλέπουν συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμογής σε περίοδο επταετίας. Και αυτό βέβαια επιτρέπει στις χώρες δικαιούχους να έχουν μια μεγαλύτερη κυριότητα των μεταρρυθμίσεων αυτών και των σχετικών πολιτικών. Βέβαια βρισκόμαστε στο ίμιση του δεύτερου αυτού μηχανισμού προνταξιακής βοήθειας και περιμένουμε να δούμε ήδη τον ερχόμενο Δεκέμβριο ποια θα είναι η επίσημη ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, μια έκθεση που δημοσιεύθηκε πέρσι και που είχε ως τίτλο η προνταξιακή συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό το οποίο λέει η έκθεση είναι ότι εν γέννη η διοικητική ικανότητα των Δυτικών Βαλκανίων δεν βελτιώθηκε και αυτό οφείλεται στην έλλειψη πολιτική βούληση από τι κυβερνήσει των Δυτικών Βαλκανίων. Λέγεται επίση στην έκθεση αυτή ότι υφίσταται ένα ακόμα λόγο ο οποίο είναι, και παραθέτω εδώ πέρα, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά δύναμη τελικά στην προσπάθειά τη να επιβάλλει μεταρρυθμίσει και αυτό ακριβώ επειδή οι μεταρρυθμίσει αυτέ δεν γίνονται στο πλαίσιο επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα-δύο για παράδειγμα, τα οποία έχουν κάνει θετικές δηλώσεις για ορισμένες κυβερνήσεις χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες κατάφορα αγνοούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, επικεφαλής των οποίων πολλές φορές είναι άτομα τα οποία βρίσκονται υπό ποινική δίωξη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αμαυρώνει πάρα πολύ την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες αυτές. Νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της οπισθοδρόμησης που έχουμε στις μεταρρυθμίσεις. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο να ξεκινήσουμε μια επίσημη διαδικασία αναλυτικής εξέτασης και ενταξιακών διαπραγματεύσεων, επιμένοντας κυρίως στα κεφάλαια 23 και 24 της ενταξιακής ε, διαδικασίας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα ε, αναγκάσουμε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να εργαστούν στο πλαίσιο ενό ε, αυστηρού πλαισίου ενταξιακών διαπραγματεύσεων και να εφαρμόσουν πραγματικά στην πράξη τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες νομοθετούν. Κατά αυτόν τον τρόπο μόνο θα υπάρχει αποτελεσματική χρησιμοποίηση του μηχανισμού προταξιακής βοήθειας. Πολύ σύντομα να αναφερθώ σε δύο επιμέρους στοιχεία. Στα πλαίσια του πρώτου μηχανισμού πρωταξιακής βοήθειας δεν υπήρχε αρκετή χρηματοδότηση για το κράτος δικαίου. Τώρα ως προς αυτό έχει βελτιωθεί η κατάσταση, στα πλαίσια δηλαδή του δεύτερου μηχανισμού πρωταξιακής βοήθειας. Έχουμε δει κάποιες θετικές εξελίξεις στην ε, όλη αυτή περιφέρεια και θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κονδύλια όσον αφορά την τι μεταρρυθμίσει για το κράτο δικαίου, μολονότι είδαμε μια σημαντική επιδείνωση. Πάλι να αναφέρω κάτι που αναφέρεται στην ειδική ε, έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Λέγεται στην έκθεση αυτή ότι τα ελεύθερα μέσα ενημέρωση και μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά το ζήτημα της διαφθοράς και του οργανωσμένου εγκλήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να στηρίξουμε την ε, κοινωνία των πολιτών και επίσης να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και επίση να καταφέρουμε να ασκούμε πίεση κάθε φορά που υπάρχει παραβίαση τη ελεύθερη έκφραση και τη ελεύθερη λειτουργία των μέσων μαζική ενημέρωση και πολλά άλλα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πέρα από αυτά τα οποία κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι πολλές φορές όταν κάνουμε δηλώσεις υπέρ της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης δεν εισακόμεθα αρκετά επιτόπου. Ας συνεργαστούμε περισσότερο με τον ΟΑΣΕ για παράδειγμα και ας χρησιμοποιήσουμε τη δική του εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύσουμε την ελευθερία έκφρασης των μέσων ενημέρωσης. Πολλά από τα αισθήματα αυτά που έχουν να κάνουν με το κράτο δικαίου και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων αποτελούν αντικείμενο πολιτικού διαλόγου με τι εμπλεκόμενε χώρε. Αναφέρομαι εδώ πέρα στον διάλογο υψηλού επίπεδου που έχουμε με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Μακεδονία, λέει ο Στην τελευταία αυτή περίπτωση, βέβαια, ο διάλογο αυτό επισκιάστηκε από την πολιτική συμφωνία του 2015 που είχε στόχο να επιλύσει την πολιτική κρίση στη χώρα αυτή. Όταν όμως ο διάλογος αυτός να οδηγεί στα αναμενόμενα αποτέλεσμα ή όπως έγινε στην περίπτωση της πολιτικής συμφωνίας με τη Μακεδονία, οι συστάσεις για ανάληψη δράσης τελικά δεν ακολουθήθηκαν με συγκεκριμένες δράσεις, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι άμεσος αρνητικός αντίκτυπος για τα προγράμματα εκείνα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλά με τρόπο στεναρό και ηχηρό κάθε φορά που δεν τηρούνται οι δεσμεύσει των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Διαφορετικά δίνουμε την εντύπωση ότι υπάρχει ένα γενικότερο καθεστώ ατιμορρησία για το οποίο δεν κάνουμε απολύτω τίποτα και το οποίο έχει να κάνει πάρα πολλέ φορέ με τα κυβερνώντα κόμματα στι χώρε αυτέ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς και είναι επεμβατική πολλές φορές προκειμένου να καταφέρει να επιβάλλει την εφαρμογή όλων αυτών των υποχρεώσεων. Ένας βουλευτής από το Κοινοβούλιο της Βοσνής Ζαγοβίνης σε μια χθεσινή συνεδρίαση ρώτησε πώς διαμορφώνεται η κοινωνία των πολιτών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα μπορούσα να μιλήσω για την Ιρλανδία. Ξέρετε ότι, για παράδειγμα, η εφαρμογή της ερευνητική διαδικασίας στη Βόρεια Ιρλανδία δεν θα μπορούσε να είχε λάβει χώρα αν δεν είχε εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών, ιδίω όσον αφορά την περίοδο μετά το τέλος των συγκρούσεων. Δεν θα πρέπει λοιπόν να θεωρείται δεδομένη συμβολή, συμβολή της κοινωνίας των πολιτών ή σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραγωνίζεται ή απλώς θεωρητικά να προβάλλεται η κοινωνία των πολιτών χωρίς όμως στην πράξη να συμβάλλει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς επίσης και σωστά λειτουργούσε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτων χωρις ομως την πραξη να συμβαλλει ειναι πολυ σημαντικο λοιπον να εχουμε ανεξαρτητα μεσα μαζικης ενημερωσης καθως επισης και σωστα λειτουργουσε οργανωσεις της κοινωνιας των πολιτων Και θα έλεγα επίσης ότι χρειαζόμαστε υψηλότερη υποστήριξη για την κοινωνία των πολιτών αφενός, αλλά επίσης και για τις ε, πολιτικές νεολαίες, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί ε, μια νοτροπία δημοκρατίας, η οποία πολλές φορές απουσιάζει από αρκετές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα ήθελα πολύ σύντομα, πρωτού ολοκληρώσω, να αφαιρθώ σε ένα δεύτερο ζήτημα, οικονομικές εξελίξεις. Μία από τις βασικές προτεραιότητες εδώ πέρα είναι να αντιμετωπίσουμε τα παράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας, 20% στη Σερβία, 29% στη Μακεδονία και πάνω από 50% της ενεργείας αυτής ε, έχει να κάνει με τους νέους. Και ξέρω ότι το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Στα πλαίσια του μηχανισμού προταξιακής βοήθειας έχει αναλυφθεί δράση προκειμένου να προωθηθεί περισσότερο η εκπαίδευση και η ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις περισσότερες χώρες όμως των Δυτικών Βαλκανίων το εκπαιδευτικό σύστημα δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ενώ σε χώρες όπως η Σερβία βλέπουμε ότι η πρόορη κατάληψη του σχολείου φτάνει το ποσοστό του 30%. Προγράμματα λοιπόν επαγγελματικής κατάρτισης είναι απαραίτητα προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα αυτό το οποίο υπάρχει μεταξύ πραγματικών αναγκών στην οικονομία και ε, προσόντων που δίδονται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Νομίζω επίση ότι θα πρέπει να δοθεί μια σημαντικότερη οικονομική υποστήριξη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και α μην ξεχνάμε ότι στα Δυτικά Βαλκάνια έχουμε πάρα πολλέ φορέ να κάνουμε χώρε οι οποίε βγαίνουν από συγκρούσει. Και για να παραθέσω ένα τον Έσον Μαλντέλα, ο οποίος αποτελεί πραγματικό παράδειγμα ηθικής ακαιρεότητας και καθοδήγησης για μας, η εκπαίδευση παραμένει ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην οικοδόμηση ενό έθνου. Αυτό είχε πει ο Νέσον Μαντέλα. Επίση, το ζήτημα τη επικοινωνία και τη ενημέρωση είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με επιτυχία προ τα έξω τα βασικά επιτεύγματά τη στον τομέα τη εξωτερική πολιτική και στον τομέα τη διεύρυνση. Βέβαια, αυτό πολλέ φορέ έχει να κάνει με την ίδια τη στάση επιμέρους κρατών μελών, τα οποία διστάζουν να μιλήσουν θετικά εσωτερικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θεωρούν ότι θα απομακρύνουν κατά αυτόν τον τρόπο ψηφοφόρου. Και δυστυχώς το ζήτημα της διεύρυνσης εμπλέκεται στα πλαίσια ενός πολύ, ε, μιας πολύ τοξικής συζήτησης αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Θεωρώ πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που τους δίνεται προκειμένου να δείξει πώς η χρηματοδότηση των Δυτικών Βαλκανίων έχει συμβάλει τελικά στο να βοηθήσει τις χώρες αυτές. Και αυτό σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σας είπα, δεν είναι ο μόνο σημαντικός διεθνής παράγοντας στην περιοχή. Για παράδειγμα, στη Σερβία υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι η Ρωσία είναι τελικά αυτή η οποία παρέχει σημαντικότερη οικονομική υποστήριξη, ενώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. Μολονότι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει να βελτιώσει τα εργαλεία επικοινωνία τη. παρόλα αυτά, θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα ακόμα, προκειμένου να δείξει ότι όντω συμβάλλει έμπρακτα στην ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Thank ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους τρεις προσκεκλημένους μας. Τώρα να σας δώσω τον λόγο για να κάνετε ερωτήσεις. Ε, προτείνω λοιπόν να ακούμε μία φορά κάποιον από τα Δυτικά Βαλκάνια και μία φορά κάποιον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε τα πρώτα ε, Να σας παρακαλέσω πρώτα να συστήνεστε και όταν απευθύνεστε σε κάποιον συγκεκριμένο από το πάνω μας, να το λέτε, ξεκινάμε με έναν γνωστό, γνωστό μας, τον κύριο Νίκολα Ποπόσκι, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, της Εθνοσυνέλευσης της Σκοπιά. Ε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Τρεις συστάσεις ε, θα είχα να κάνω και προς την Κομισιόν και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς περνάμε από το ΕΠΑ στο ΕΠΑ 2 και τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση πρώτων. Θεωρώ ότι στο ΕΠΑ 2 ο ανταγωνισμός είναι καλός και πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το στοιχείο και μεταξύ κλάδων, ε, γεωργία, υποδομές κτλ μεταξύ φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και κρατών και μεταξύ χωρών. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο, το αποτελεσματικότερο μέσο είναι η πίεση από τους άλλους. Δεν πρέπει να το αποκλείουμε, θα μας βοηθήσει και θα βοηθήσει και σας βεβαίως να δικαιολογήσετε το πώς ξοδεύετε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Το δεύτερο, η αξιολόγηση από εξωτερικούς αξιολογητές. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί φεύγει έτσι θα έλεγα η οπτική γωνία της διοίκησης της ε, Βρυξέλλες. Αλλά είναι ύποπτο γιατί υπάρχει η υποψία της πελατειακής σχέσης. Τη στιγμή που βασίζεται μόνο σε εξωτερικούς αξιολογητές μπορεί να θελήσουν να σας ικανοποιήσουν και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και ε, έχουμε και το θέμα της πολιτικής αξιολόγησης αυτό, το οποίο λοιπόν είναι λογικό να στηριχθεί η περιοχή μας το τρίτο στοιχείο, μια που μιλάμε για πολιτικές προτεραιότητες, πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η ένταξη περιφερειακή εμείς. Έχουμε αλληλεγγύα στο να λέμε ότι η Ευρώπη προσπαθεί να ανασυστήσει την πρώην ε, Ομοσπονδία της Ιουγκοσλαβίας, ειδικά όταν έρχεστε στη χώρα μας και καμιά φορά μας το λέτε κιόλα, μας λέτε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, ε, αλλά πρέπει να ενταχθούμε. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να έχουμε έναν ελεύθερο χώρο, να ταξιδεύουμε ελεύθερα, ε, να ενταχθούμε στο roaming, ευκολότερη πρόσβαση. Είναι ευκολότερο να πάει κανείς από το Σκόπια στις ε, Βρυξέλλες παρά στο Σεράγεβο. Ενώ βεβαίω η απόσταση δεν συγκρίνεται. Η οικονομία ε, Επίση λέει τα πάντα και αυτό ελπίζουν και οι δικοί μα οι φορολογούμενοι είμαστε μία από τι πιο ανοιχτέ οικονομίε μα. 70% των εμπορικών μα σχέσεων είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% είναι με τις χώρες που λέτε εσεί Δυτικά Βαλκάνια αυτό πρέπει να εξελιχθεί σε τον χρόνο και τέλο. πρέπει να υπάρξει μία μετατόπιση προς ε, περισσότερες υποδομές για να βοηθηθεί η πρόσβαση στην περιοχή και λιγότερη δημόσια διοίκηση. Εξακολουθούν στα Βαλκάνια να πηγαίνουν οι ικανοί στην ε, διοίκηση. Αν είσαι πραγματικά καλό σε δυτικέ χώρε, υπάρχουν δυσκολίε να πάει κανεί στη δημόσια διοίκηση. Στι δικέ μα ε, γίνεται αυτό. Αν είσαι πολύ πραγματικά καλό, πηγαίνει να δουλεύει στη Γερμανία. Αλλά εξακολουθούμε να έχουμε ικανού ανθρώπου που είναι στην διοίκηση. Οπότε λιγότερα λεφτά στην διοίκηση και περισσότερα λεφτά στις υποδομές μεταξύ των πόλεων μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Νίκολα. Λέτε ότι εμείς λέμε την περιοχή Δυτικά Βαλκάνια. Ξέρω πως δεν σας αρέσει. Αν δεν έχει βρεθεί ακόμα μια καλύτερη ονομασία. μπορούμε να πούμε και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτά λοιπόν, να τα έχει υπόψη της η γραμματεία. Α, νομίζω ότι το σημειώσαμε. Ο κ. κατόπιν από τους σοσιαλδημοκράτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαρίτια Σχάκε γιατί θεωρώ πως υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα εδώ δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι για το πώς ε, έχουν χρησιμοποιηθεί τα μέσα αυτά μέχρι Όχι ότι είναι όλα λάθος, αλλά παρατηρούμε κάποια πράγματα. Ο κόσμος στις χώρες αυτές, και εγώ δεν μπορώ να λέω Δυτικά Βαλκάνια είναι αστείο, πρέπει να σημειώσουν λοιπόν ότι και στις δύο πλευρές εργαζόμαστε εντατικά για να ανοίξουμε το δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό πρέπει να προσέξουν να γίνουν οι σωστές μεταρρυθμίσεις και να αλλάξει η ζωή τους θετικά. Πρέπει να παρατηρήσουν και ε, να προσέξουν ότι και η ασφάλεια αυξάνεται μέσω της σταθερότητας, αλλά κατά τα λοιπά το θέμα αφορά την βοήθεια στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για να δείξουμε ότι πραγματικά τους θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σημαίνει όχι μόνο να δώσουμε λεφτά για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και σύμβουλων αλλά και για υποδομές υπό το σκοπιά της ένταξης αντίστοιχα για αυτό το οποίο ε, λέμε την ανταλλαγή νέων ε, επαφών κτλ. Και βεβαίω, εντάξει, δεν να αυτά ξαφνικά, αλλά δεν φαίνεται κάτι. Γιατί δίνουμε και το τελευταίο send και μετά δεν έχουμε 20 ευρώ για τη γνωστή αυτή πινακίδα ε, έργο χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να δούμε το θέμα αυτό της ολοκλήρωσης γιατί δεν ικανοποιεί και κάποιες κυβερνήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και είπατε ότι δεν είναι μόνο η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία και άλλες χώρες που ενδιαφέρονται για να αυξήσουν την επιρροή τους. Όποιο θέλει οπωσδήποτε να συνεργαστεί με τη Ρωσία μπορεί να το κάνει, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες. Η Σαουδική Αραβία που εμπλέκονται πολύ. Πρώτο τελευταίο θέμα. Θεωρώ ότι Πρέπει να φύγουμε από την σκέψη ότι το άνοιγμα ενός κεφαλαίου είναι κάτι το επαναστατικό για τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα. Ξέρουμε ότι είναι αναγκαίο και σημαντικό, αλλά ένας φούρναρης ε, εκεί πέρα στο Βελιγράδι δεν θα στολίσει το μαγαζί όταν ακούσει ότι ανοίξαμε δύο κεφάλαια Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Και θεωρώ ότι το τελευταίο αυτό πράγμα που είχαν οι άνθρωποι ήταν η απελευθέρωση της ε, βίζας. Δυστυχώς όχι το κοσφοπέδιο όπου ε, χτες ε, ζητήσαμε από την Κομισιόν να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Αλλά Ίσως η συμπερίληψη στο ευρωπαϊκό σύστημα roaming να ήταν ε, ένα θέμα, κάτι το απτό που θα το παρατηρούν όλοι. Οι νέοι ε, και οι επιχειρηματίε ε, στις πόλεις, Η μία πόλη και στην άλλη. Τελευταίο. More for more. Ε, το λέμε έτσι γρήγορα, αλλά πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Πρέπει να μπορούμε να είμαστε κάπως πιο ενεργοί σε αυτά τα θέματα και συγκεκριμένα όσον αφορά τα μέτρα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προτεκτοράτα, θέλουμε εταίρους. Και αυτό γίνεται μόνο με διάλογο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κνούτ Φλέκενστάιν. Το επόμενο επόμενος ομιλητής είναι ο Φάντιο Σεντέλη από την Μακεδονία από την ομάδα το κόμμα Μπέζα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ε, Κοινοβουλίων των Δυτικών ε, Βαλκανίων, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των κονδυλίων από το μηχανισμό προνταξιακής βοήθειας. Θα ήθελα να αφαιρθώ λοιπόν στο σύστημα ελέγχου όσον αφορά τη χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων, καθώς επίσης και σε ένα άλλο μέσο που έχει να κάνει με την αξιολόγηση του επίπεδου διαβίωσης. Αναφερόμαστε σε ένα σύστημα ελέγχου που έχει να κάνει με τα κοινοτικά κονδύλια. Πολλέ φορέ όμω δεν καταφέρνουμε εμεί οι ίδιοι να ελέγξουμε σωστά τα του δικού μα εγχώριου προπολογισμού. και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ε, εμπλέκονται όλο και περισσότερα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των ε, κοινοτικών κονδυλίων σε διάφορες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όπως και στη δική μου τη χώρα, την ε, Μακεδονία. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική χρησιμοποίηση των κονδυλίων αυτών και θα πρέπει προφανώς να διοχετεύονται στους σωστούς δικαιούχους και να μην συμβάλλουν απλώς στον καταφέρνουν οι κυβερνήσεις να επιβιώνουν ή να τα βγάζουν πέρα δημοσιονομικά. Στόχος του κονδυλίου αυτών, όπως είπατε, είναι οι χώρες του Δυτικών Βαλκανιού να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γενικότερη τάση στις χώρες μας όμως είναι ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να έρθουμε όντως πιο κοντά σε εσά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μερικές φορές πρέπει να σας ξεκαθαρίζουμε κάθε φορά ότι πρέπει να είναι αμοιβαία και αμφίδρομη διαδικασία αυτή και εμείς να έρθουμε πιο κοντά σε εσά αλλά και εσείς προς εμάς. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Χρειαζόμαστε και Ευρωπαίου αξιωματούχου που να έρχονται στι δικέ μα χώρε, αλλά και αξιωματούχοι από τι δικέ μα χώρε να εκπαιδεύονται σε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Σόλτε το έχει το λόγο από του Πρασίνου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Τα κονδύλια αυτά από το Μηχανισμό Προταξική Βοήθεια είναι πολύ σημαντικά για την ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Αναφερόμαστε όλο και περισσότερο για τον αναλυτικό έλεγχο που θα πρέπει να γίνεται για τη χρήση των κονδυλίων αυτών και λέμε επίση ότι θα πρέπει να έχουμε εξωτερικά όργανα που να κάνουν τον έλεγχο αυτό, πέρα από του εσωτερικού δηλαδή ελέγχου που θα πρέπει να γίνουν. Πάντως, κάθε μία από τις χώρες αυτές στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων έχει τις δικές της εσωτερικές ελεγκτικές αρχές. Οι αρχές λοιπόν αυτές θα πρέπει να δραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της επαλήθευσης και του ελέγχου της χρησιμοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων. Πέρα από αυτό όμως πρέπει να απαντήσουμε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Δεν είναι σημαντικό μόνο να βλέπουμε ποια είναι η πορεία των κονδυλίων αυτών και αν όντως χρησιμοποιούνται με έναν τρόπο αξιόπιστο. Πρέπει επίση να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά του, την αποδοτικότητά του και αν μπορούμε να οδηγηθούμε και σε μια κάποια εξοικονόμηση. Νομίζω ότι και το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα κράτη-μέλη. Πώς μπορούν να καταμετρήσουν τελικά και να αποτιμήσουν την απόδοση των κονδυλίων αυτών. Το θέμα δεν είναι να δαπανά κανεί μόνο τα κονδύλια αυτά, αλλά να μπορεί να είναι και υπόλογο για τον τρόπο που ε, δαπανώνται αυτά τα κονδύλια και τελικά ποιο είναι ο αντίκτυπο των κονδυλίων αυτών για διάφορε πολιτικέ, για τη ζωή των πολιτών, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και κ.ο.κ. Θα μπορούσα να συμφωνήσω με του προσλαλήσαντε ότι όντω η υποδομή είναι πολύ σημαντική, η διασύνδεση μεταξύ των χωρών τη ε, περιοχή αυτή, αλλά Εξίσου σημαντικό είναι να δούμε πώς οι χώρες του Δυτικών Βαλκανίων εφαρμόζουν την εγκριθήσα νομοθεσία. Εκ πρώτης όψεως θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι περισσότερες χώρες του Δυτικών Βαλκανίων έχουν πλέον ένα νομοθετικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο μάλλον, το οποίο συνάδει με το ενωσιακό κεκτημένο αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι δεν καταφέρνουν πολλές χώρες να εφαρμόσουν σωστά την νομοθεσία αυτή. Εκεί υπάρχουν αρκετές αδυναμίες. Πρέπει λοιπόν να επενδυθούν κάποια κοινοτικά κονδύλια από το μηχανισμό προταξιακής βοήθειας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν προγράμματα κατάρτισης για αξιωματούχους του δημοσίου τομέα, για καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών που απορρέουν από τα κονδύλια αυτά και για να υπάρχει ένας υψηλότερος βαθμός διαφάνειας. Νομίζω λοιπόν ότι και οι βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν ώστε να παρακολουθούμε καλύτερα τη χρήση των κονδυλίων αυτών. Ευχαριστούμε τον Ίγκορ Σόλτες. Δύο ακόμα έχουν ζητήσει το λόγο από το Κωσυφοπέδιο αυτή τη φορά. Ο κύριος Αμπτούλα Χώτη πρώτος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο floor is yours. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά συμμετέχω στο φόρουμ αυτό και θα σας δώσω την άποψή μου ως μέλος της κυβέρνησης Υπουργός Οικονομικών και μέλος της ομάδας σχεδιασμού σχετικά με τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων IPA. Θα μιλήσω καταρχάς για την ε, υλοποίηση των πόρων IPA. Κατά την άποψή μου πρέπει να αφιερώσουμε πολύ περισσότερο χρόνο στο σχεδιασμό και στον συντονισμό με την κυβέρνηση ώστε οι στόχοι IPA να υλοποιηθούν πλήρως. Θα πρέπει όμως να συμμετάσχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς από πρώιμο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στην ενίσχυση της κυβερνικής δυνατότητας όχι μόνο στην εφαρμογή IPA αλλά και στη δημιουργία μακροπρόθεσμου δυναμικού δυνατότητος ώστε να ακολουθηθεί μακροπρόθεσμα η κατεύθυνση που υποδεικνύει το πρόγραμμα IPA. Και ως πρώην Υπουργό Οικονομικών, σκιώδης αν θέλετε Υπουργός Οικονομικών, ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε τις δυνατότητες μας. Χρειάζεται συγχρηματοδότηση αυτής της προσπάθειας. Τώρα για τα ίδια τα προγράμματα IPA έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους ε, και ε, κάποια, ε, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε την αίσθηση ότι χάνουμε την όθηση Και λόγω των καθυστερήσεων αυτών δημιουργείται ένα κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης από τους ε, πολίτες. Θα πρέπει να μείνουμε στις κατευθυντήριες γραμμές ώστε να έχουμε το ευκταίο αποτέλεσμα. Ε, τεχνικός μιλώντας, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η χρηματοδότηση IPA είναι, ναι, χρηματική στήριξη προς τις χώρες αυτές, οικονομική στήριξη, αλλά είναι και μια πολιτική χειρονομία. Και ίσως θα έπρεπε να δίνεται περισσότερη έμφαση στο στοιχείο αυτό, στην πτυχή αυτή, να δημοσιοποιείται δηλαδή εμφανέστερα και να δίνεται και η δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να ελέγχει την πορεία του προγράμματος. Προφανώς και μου φαίνεται και εμένα θετικό το γεγονός της εξωτερικής ανεξάρτητης αξιολόγησης, αλλά και οι εσωτερικοί θεσμοί της χώρας θα πρέπει να δουν την χρησιμοποίηση των πόρων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει συνολικά να είναι εμφανέστερη στην όλη περιοχή, ώστε να είναι προφανές για τους πολίτες πώς δαπανώνται, πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι αυτοί. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σόλε τώρα, εισηγητής ε, των Πρασίνων για τον IPA. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο έχω ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Όπως ακούσαμε από τους ομιλητές και όπως γνωρίζουμε από την ε, εμπειρία μας ε, της υλοποίησης ε, των κονδυλίων IPA, η απόδοση σχετίζεται με διάφορους παράγοντες. Καταρχάς, με την πολιτική βούληση των δικαιούχων. Και δεύτερον, με τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πιέσει και να απαιτήσει πραγματικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές. Τώρα, κάποιες φορές σημειώνεται ένα έλλειμμα, αν θέλετε, πραγματικής πολιτικής βουλήσεως να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις Ε, και κάποιες φορές επίσης περιορίζεται και η δυνατότητα ή η, βόληση, η η βουληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πιέσει προς την κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων αυτών. Δεδομένων των δύο αυτών περιορισμών θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να αναγνωριστούν και να υπογραμμιστούν. Χρειάζεται λοιπόν η στήριξη αφενός της κοινωνίας των πολιτών η οποία μπορεί να είναι ένας πραγματικός παράγοντας αλλαγής σε κάθε κοινωνία, αλλά και βεβαίως και στις χώρες για τις οποίες μιλούμε. Και δεύτερον, το σύστημα επιβράβευσης. Και περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον ε, την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος αυτούς συστήματος αυτού, με συγχωρείτε, επιβράβευσης. Ακούσαμε τώρα από τον συνάδελφο από την Μακεδονία ένα στοιχείο σχετικά με την περιφερειακή ολοκλήρωση και την τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη που θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση αυτήν. Η ερώτηση είναι τα προγράμματα, τα πολυμερή που αφορούν σε πολλές χώρες δηλαδή του IPA θα μπορούσαν θεωρείται να βοηθήσουν προς αυτήν την περιφερειακή ολοκλήρωση. Η ερώτηση αυτή απευθύνεται κυρίως στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Σόλε. Νομίζω ότι έχουμε άλλον έναν ομιλητή και μετά θα ήθελα να κλείσω τον κατάλογο γιατί θέλουμε να ακούσουμε τα μέλη του πάνελ. Μέμλη Κρασνίκη από το Κοσυφοπέδιο λοιπόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος διότι πιστεύω ότι ο κύριος Χώτη κάλυψε τα ουσιαστικά στοιχεία της ε, εμπειρίας χρησιμοποίησης των πόρων IPA στο Κόσοβο. Καταρχά να πω ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέσο. Έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε μερικές από τις περιοχές υψηλότητα της προτεραιότητας για τη χώρα. Μέσω της άμεσης εμπειρίας που είχα ως υπουργό στις προηγούμενες δύο εντολές πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του την αποτελεσματικότητα υλοποίησης του ίδιου του μέσου. Πριν από δύο μήνες στο Κόσοβο το IPA 2014 ξεκίνησε, επομένως με τριετή καθυστέρηση. Είμαστε ήδη στην ενδιάμεση επανεξέταση αλλά μόλις ξεκίνησε το IPA2. Θα χρειαστούν δύο χρόνια για τις συμβάσεις αυτές και επομένως θα ολοκληρωθεί το IPA 2014 κάπου προς το 2020, στο τελευταίο έτος του IPA. Επομένως η αποτελεσματικότητα είναι ε, όρος κλειδί, διότι αυτή ήταν η εμπειρία που είχαμε νομίζω σε όλες τις χώρες της περιοχής καθυστερήσεις, γραφειοκρατικές διαδικασίες, το οποίο σε κάποιο βαθμό κατανοούμε, αλλά θα χρειαστεί να έχουμε μια συζήτηση για το πώς θα γίνει η όλη διαδικασία ομαλότερη και ταχύτερη. Τώρα, επιδόσεις. Ακόμα και όταν τα προγράμματα ξεκινήσουν να υλοποιούνται, χρειάζεται πρόσθετος χρόνος, συνήθως. Κάποια από τα έργα που υλοποιούνται στο Κόσοβο έχουν μια αρχική πρόβλεψη δεκαοκτάμινη ή διετή. Αλλά συνήθως δίνεται μια παράταση, γίνεται μια καθυστέρηση τουλάχιστον ενός έτους, γιατί όλα περιπλέκονται. Η αποτελεσματικότητα, δηλαδή το πόσο εύχριστα είναι τα προγράμματα στο ε, πεδίο, στο έδαφος. Έχουμε success stories, αλλά έχουμε και εμπειρίες περιορισμένης επιτυχίας. Υπήρχε αρκετό υλικό τεχνικής βοήθειας, το οποίο όμως τελικά δεν έφτασε στον προορισμό του. Και αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα μεταξύ των δικαιούχων, των κυβερνητικών φορέων, γιατί δυστυχώς θα μπορούσαμε να γεμίσουμε μια αίθουσα με επιτυχείς εκθέσεις και έγγραφα τα οποία όμως δεν χρησιμοποιούνται δυστυχώς από τόσο πολυάριθμους δικαιούχους. Η χρησιμότητα λοιπόν, το εύχριστο των προγραμμάτων αυτών είναι ένα θέμα. Στις κεφαλαιακές επενδύσεις η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική. Χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ της τεχνικής αρρωγής και των δαπανών. Ε, στο Κόσοβο είχαμε, στην Μητρόβιτσα, είχαμε χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό αθλητικό πρόγραμμα ώστε να το εκμεταλλευτεί η τοπική κοινότητα, οι νέοι και λιγότερο βασιστήκαμε στην τεχνική βοήθεια, αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχει αυτή η λογική της κατανομής των πόρων. Χρειάζονται αμοιβέ για τους ε, συμβούλους, ε, χρειάζεται TA, χρειάζονται έργα ολοκλήρωσης ή τελειοποίησης κάποιων εγγράφων. Και τέλος να πω επίσης ότι ο σχεδιασμός όπως και η επανεξέταση, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις προτεραιότητες των δικαιούχων. Πρέπει να ταιριάσουμε τις δαπάνες, τα κονδύλια με τις πολιτικές προτεραιότητες, αλλά δεν είναι πάντα ταιριασμένα αυτά. Άλλο ένα παράδειγμα από το IPA2, γεωργική ανάπτυξη στο Κόσοβο, μία από τις τρεις βασικές περιοχές, δεν είναι πλέον περιοχή προτεραιότητας. Ποιος έλαβε την απόφαση, δεν είμαι βέβαιος, εγώ ήμουν υπουργό Γεωργίας. Εγώ δεν έλαβα την απόφαση και ούτε με ρώτησε κανείς Επομένως, το πρόβλημα που δημιουργείται κατά τον τρόπο αυτόν γίνεται ένας μακροπρόθεσμος ε, σχεδιασμό για το 14-20, λαμβάνοντα υπόψη τους πόρου που έχουν αφιερωθεί στον IPA από την αρχή. Όμως όταν αλλάξουμε τη στόχευση αυτό επηρεάζει και, τις, ε, και τον ενδιάμεσο σχεδιασμό της ίδιας της χώρας. Εάν οι δικαιούχοι δεν έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία της οποιασδήποτε επανεξέτασης ή αναθεώρησης, τουλάχιστον σε υψηλό επίπεδο, γιατί μπορεί να συμμετέχουν κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί ε, μέσου επίπεδου, αλλά χρειάζεται το υψηλότερο επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Και υπάρχουν και διαφορά απόψεων ακόμα και στις ε, Βρυξέλλες σε σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη γεωργική ανάπτυξη. Πολύ διαφορετικές απόψεις εκφράζονται από την γάμα δελτα νίρ και τη γάμα δελτα άγκρη. Επομένως, εσείς θεωρείτε ότι δεν θα ήταν σημαντικό να συμπεριλάβουμε στο σχεδιασμό αυτών οπωσδήποτε τους δικαιούχους αλλά και τις υπόλοιπες γενικές διευθύνσεις που ασχολούνται με τους συγκεκριμένους τομείς επί του συγκεκριμένου που μόλις ανέφερα η ΓΑΜΑ Άγκρη όπου έχουν την ανάλογη εμπειρία και τη δυνατότητα να ασχοληθούν με αυτά τα στοιχεία περισσότερο ίσως από τη Γαμαδελτανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τελειώνει εδώ ο κατάλογος των ομιλητών και θα δώσω τον λόγο στους ε, τρεις πανελίστες μας ξεκινήσω πάλι με την Μαρίτια Σχάκη και μετά θα συνεχίσουμε με την κυρία Καλαβέρα και τον κύριο Φουέρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και για τις ειλικρινείς ε, παρατηρήσεις σας, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτό το οποίο λοιπόν βγάζω ως συμπέρασμα είναι ότι ουσιαστικά η φιλοδοξία υπάρχει. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε. Όσον αφορά τώρα τις πιο αποτελεσματικές δαπάνες, την επικοινωνία, αλλά και τις ξένες επιρροές από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω αυτά είναι τα βασικά τα οποία προέκυψαν. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα ακριβώς ε, της ε, πολιτικής δέσμευσης και αυτό σημαίνει υπεύθυνη διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι πολύ λεπτό το θέμα αυτό της ένταξης και των σχετικών κονδυλίων. Γιατί δεν μιλάμε για αναπτυξιακή βοήθεια, τα μέτρα αυτά σημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρξουν ψηλότερε προδιαγραφέ για το κράτο δικαίου, κοινωνία των πολιτών, οικονομική ανάπτυξη, ελευθερία των ΜΜΕ και περιφερειακή ολοκλήρωση. Και δεν είμαι σίγουρος, ε, σίγουρη ότι γίνεται αντιληπτό. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική η σχέση μεταξύ όλων των διαφορετικών στοιχείων που είναι μέρος της διαδικασίας εφαρμογής από την ενίσχυση των θεσμών, στην καταπολέμηση της διαφθοράς, την βελτίωση της εποπτείας που μετά βεβαίως με τη σειρά της θα βελτιώσει την ικανότητα να εφαρμόσουμε σωστά την προενταξιακή βοήθεια. Όχι μόνο λοιπόν απομονωμένα ως οικονομική ανάπτυξη, αλλά για να ενισχυθεί η δημοκρατία και η κοινωνία γενικώ. Και τέλος, και ως βουλευτές αυτό είναι πάντα πρώτη μας προτεραιότητα και πρέπει να είναι σαφές ότι εμείς βεβαίω θέλουμε να καλωσορίζουμε και να ε, υπάρχει ακριβώς η ευημερία του κόσμου δεν είναι κάποιο τρόπο για να αρπάξει κάποια κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να καταλήγει σε αυτούς οι οποίοι το χρειάζονται. Και υπ' αυτό το πρίσμα, και αυτό το απευθύνω περισσότερο σε αυτούς που εργάζονται στον στρατηγικό διάλογο, υπ' αυτό το πρίσμα θα τα δει τα θέματα το Κοινοβούλιο, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ψηλή προτεραιότητα και σημαντικό για να μπουν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα οικοδομηθούν όλα τα άλλα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία να έχουμε αυτήν την συνάντηση και ελπίζω να είμαστε σε επαφή και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ Μαρίτια. Κυρία Ρουίς Καλαβέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία Σάκε. Να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς σας Ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούει τις απόψεις σας, όχι μόνο σήμερα προφανώς. Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί σας και με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου η ενδιάμεση αναθεώρηση να εμπλουτιστεί πραγματικά από την πραγματικότητα που ισχύει επί τόπου. Κάποιες σκέψεις κοινωνία των πολιτών, πάρα πολύ σημαντική σίγουρα και όχι μόνο ως προς τη χρηματοδότηση. Χρηματοδοτούμε μέσω κονδυλίων προγράμματα που στηρίζουν ε, την κοινωνία των πολιτών και τα σχετικά δίκτυα, αλλά είναι πολύ σημαντικό και σε επίπεδο κοινοβουλίου, δηλαδή τα κοινοβούλια κάθε φορά που επεξεργάζονται νέα νομοσχέδια είναι σημαντικό να κάνετε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών. Προκύπτουν ε, συχνά καταστάσεις όπου τελικά προχωρούμε στα κοινοβούλια με διαδικασία του fast track χωρίς να γίνεται διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι ο δικός σας ο ρόλος θα εμπλέκει και την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει λοιπόν μέσω της απαραίτητης διαβούλευσης να ακούτε και την κοινωνία των πολιτών. Δεύτερον, σίγουρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και συμφωνώ εδώ πέρα με τον Νικόλα Ποπόσκι, όπου η γενικότερη αυτή περιφέρεια έχει καταβάλει πάρα πολλές προσπάθειες ε, τα τελευταία χρόνια προκειμένου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να στηριχθεί και αυτό θα γίνει μέσω και των πολυκρατικών διακρατικών αυτών προγραμμάτων που έχουμε. Προφανώς όλοι ενδιαφερόμαστε να ενισχύσουμε τις υποδομές της περιοχής αυτής. Πρέπει να συνδεθεί η περιοχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι επιμέρους χώρες περιοχής μεταξύ τους. Πρέπει όμω να ξέρουμε ότι από, μόνες, από μόνη τη η ενίσχυση υποδομή δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση. Όσου αυτοκινητοδρόμους και να δημιουργήσουμε, αν δεν εναρμονίσετε την πολιτική σα στους συνοριακούς ελέγχους δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση για τα φορτηγά θα συνεχίσει να υφίσταται. Οι επενδύσεις λοιπόν θα πρέπει να συνοδεύονται με μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις προκειμένου να τροποποιηθούν οι κανονισμοί σα όσον αφορά τι οδικέ μεταφορέ εν προκειμένου. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε σε περιφερειακό επίπεδο τι μπορείτε να κάνετε, πώ μπορείτε δηλαδή να προχωρήσετε σε μεγαλύτερη περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση και ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πρωθυπουργοί που συνεδρίαση που έγινε στην Τεργέστη πέρυσι είχαν δεσμευτεί για μια τέτοια ενισχυμένη περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία. Ένα τρίτο τώρα μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε ο ρόλος που μπορείτε να διαδραματίσετε εσείς ως κοινοβούλια, το ζήτημα του ενδελεχούς ελέγχου και συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν εδώ πέρα. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε προφανώς μηχανισμούς παρακολούθησης και εποπτείας. Αναφέρομαι σε όλους αυτές τις αποστολές εξωτερικής επιθεώρησης και ελέγχου. Έχουμε και τις δικές μας υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε και την Όλαφ, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχετε όμως και εσείς τις δικές σας εθνικές ελεγκτικές αρχές. Αυτές ακριβώς πρέπει να υποστηρίξετε, να έχουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, το απαραίτητο προσωπικό και να είναι κυρίως ανεξάρτητες αρχές σε σχέση με την επιρροή που θα μπορούσε να ασκήσει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν ο ρόλο σα είναι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να δημιουργήσετε τι απαραίτητε προποθέσει για να λειτουργούν ομαλά οι αρχέ αυτέ ελεγκτικέ. Τώρα, ο σχεδιασμό και ο προγραμματισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο σημαντικό, γιατί του το πρόγραμμα αυτό του μηχανισμού προταξιακής βοήθειας είναι ένα πολιετές πρόγραμμα. Συντοποιούμε ότι ο μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας δεν θα γίνει εν μία νυχτή. Συντοποιούμε ότι όλη η διαδικασία είναι πολιετής. Σαφώς απαιτούνται αρκετοί έλεγχοι. Κάθε φορά όμως που θέλουμε να προχωρήσουμε και στο επόμενο στάδιο, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος, είναι απαραίτητη η εφαρμογή της νομοθεσίας η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό όταν είπα στην αρχική μου παρέμβαση ότι χρειαζόμαστε μία προσέγγιση υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που να υποστηρίζεται από όλες τις πολιτικές ομάδες. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά αλλάζουν οι κυβερνήσεις στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και ξεκινάμε πάντα από το μηδέν και αυτό οδηγεί σε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και πολλές φορές ακόμα και σε κατασπατάληση των ε, χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Σε κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά για παράδειγμα τη δημόσια διοίκηση ή την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, εκεί πέρα πραγματικά θα πρέπει να εμπλέκονται όλα τα πολιτικά κόμματα, όλο το πολιτικό φάσμα των κοινοβουλίων σας. Αυτό πραγματικά πρέπει να το μεταδώσετε σαν μήνυμα όταν θα επιστρέψετε στις χώρες σας. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο, με την ε, πολυκο, πολυκομματική αυτή υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων, θα καταφέρουμε τελικά να σημειώσουμε πρόοδο στον ε, διάλογο αυτό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τώρα όσον αφορά την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική επικοινωνίας. Προβλέπονται πάλι επιμέρους κονδύλια για την πολιτική επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαν να σας περισσότερα πράγματα οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας. Ξέρετε, η επικοινωνία δεν έχει να κάνει μόνο με το να βάλουμε το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πινακίδα ή να βάζουμε τη σημαία μας εδώ και εκεί έχει να κάνει πραγματικά και με την συμμετοχή που μπορούμε να έχουμε επιτόπου συνεργαζόμενοι με τις κυβερνήσεις και τα τοπικά κοινοβούλια. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι εσείς στις δικές σας τις χώρες, οι δικές σας τοπικές αρχές να αρχίσουν να μιλάνε λίγο περισσότερο για τη θετική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε τελικά να προβάλλουμε περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θετικό της ρόλο στις χώρες σας Ιδίω όσον αφορά τον ευρωπαϊκό δρόμο των χωρών σα Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φερα έχει τώρα το λόγο, τελευταίος ομιλητής. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους όσους ε, σχολίασαν κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα η περιφερειακή συνεργασία και τα προγράμματα πολλών χώρων. Ήδη υπάρχουν πολύ σημαντικά τέτοια προγράμματα και θεσμικά όργανα πολλών χωρών όπως η μεταρρυθμίση, η σχολή ε, της δημόσιας διοίκησης στο Μαυροβούνιο, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση να χρησιμοποιηθούν αυτά τα θεσμικά όργανα, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Ειδικά όσον αφορά τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου πέρσι επεσήμανε ότι υπήρχε ελάχιστη χρησιμοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του σχολείου από μία-δύο χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Οπότε πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση εντός της χώρας έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά να έχουν αντίκτυπο. Για το θέμα της εφαρμογής και της έγκρισης της νομοθεσίας συμφωνώ εδώ με την συνάδελφο ότι δυστυχώς Έχουμε δει μια κατάσταση όπου τα κοινοβούλια της περιοχής απλά κάνουν τα τυπικά στα χαρτιά και το κοινοβούλιο εγκρίνει τη νομοθεσία που καλείται με ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν υπάρχει μια διαδικασία διαβούλευσης με τους κλάδους της κοινωνίας που επηρεάζονται από αυτήν την νομοθεσία π.χ. για την νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους που θα επηρεαστούν από αυτήν την νομοθεσία. Και δεύτερον, ο φορέας που θα εφαρμόσει αυτή την νομοθεσία πρέπει να εκπροσωπείται και να έχει και εκπροσώπους αυτόν τον κλάδο. Αλλά δυστυχώς έχουμε παραδείγματα στις εκθέσεις της Κομισιόν όπου οι φορείς αυτοί αποτελούνται από μέλη κομμάτων. Απλά. Που δεν ε, αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα των ανθρώπων που θα επηρεαστούν από την νομοθεσία. Έχουμε λοιπόν ε, ακριβώ πέρα το ότι πρέπει να τονιστεί η σημασία της συνένεσης εντός των κοινοβουλίων. Αυτά είναι νομοθετήματα τα οποία έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν, να ενισχύσουν τις ε, συνθήκε ζωής στι χώρε αυτές. Όχι επειδή το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επειδή θα ωφελήσουν τις χώρε αυτές. Αλλά για να τις ωφελήσουν πρέπει να περιλαμβάνουν μια συστηματική διαβούλευση με όλους τους φορείς της κοινωνίας έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα και τις ανάγκες της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για την διαδικασία ένταξης για τις χώρες που είναι ήδη σε αυτήν την διαδικασία. Η ανάγκη δηλαδή συνένεσης σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε η, η φωνή της χώρας να εκπροσωπεί όλους τους τομείς της κοινωνίας και όχι μόνο την κυβέρνηση ή τα πολιτικά κόμματα. Και τέλος, αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω, αυτό το οποίο είπε πρόσωπος του κόμματος Μπέσα από την Μακεδονία, ότι πολλοί από εμά έχουμε τονίσει την σημασία της κοινωνίας των πολιτών, όχι μόνο την στήριξή της από την Ένωση, αλλά και ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι ανοιχτές προς την κοινωνία των πολιτών με τρόπο που δεν θα είναι κομματικός. Και δυστυχώς είχαμε παραδείγματα ε, χρηματοδότησης από εθνικές κυβερνήσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών οργανώσεων που είναι όλες κομματικές και δεν αντικατοπτρίζουν τον ρόλο της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών που είναι δηλαδή να λογοδοτεί η κυβέρνηση. Αυτό είναι ο ρόλος τους. Και δεν πρέπει να καταδικάζονται ή να παροχλούνται. Και θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες... για στήριξη της κοινωνίας των πολιτών στο τοπικό επίπεδο. Τα έργα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία των πολιτών, ειδικά τις μικρές εκείνες οργανώσεις που δεν έχουν τους πόρους ή την τεχνογνωσία, πρόσβαση στα κοινωτικά κονδυλία. Ε, ένα σύστημα δηλαδή με το οποίο θα μπορούν να περιληφθούν γιατί όταν εργαζόμουν στις χώρες αυτές ε, και στην Νότια Αφρική και στη Λατινική Αμερική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο πάντα μου έκανε εντύπωση είναι ο μεγάλος αντίκτυπος των μικρών έργων ότι δηλαδή ενώνουν ανθρώπους από διαφορετικές κοινότητες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Μακεδονία χρηματοδοτήσαμε ένα έργο για την διδασκαλία της ιστορίας από την Επιτροπή του Ελσίνκη που βεβαίως είχε δασκάλους από τις δύο κοινότητες της χώρας για να υπάρξει μια αντικειμενική ερμηνεία της σύγκρουσης του 2001. Ήταν δύσκολο οπωσδήποτε ήταν ζητήματα έντονα, τα συναισθήματα υπάρχουν ακόμα. Επίσης ένα έργο το οποίο ανέδειξε τις προκαταλήψεις, αλλά ακριβώ αυτό ήταν το σκεπτικό. Και καταλήξαν με ένα αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα, αλλά βεβαίως εάν η κυβέρνηση δεν το α, σωματώνει στα μαθήματα του σχολείου δεν παίζει κανένα ρόλο, δεν έχει κάποιο νόημα. Είναι ένα παράδειγμα όμως μικρών έργων σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο που μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο να ενισχύσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης. στα διαφορετικά επίπεδα μεταξύ εθνικών κοινοτήτων και μεταξύ των κοινοτήτων γενικώς. Γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις ε, κοινωνιών που έχουν βγει από συγκρούσεις. Η δυσπιστία είναι μεγάλη. Και ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό, να έχουμε αυτά τα έργα και βέβαια οι καλύτερη φορείς είναι οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών στο τοπικό επίπεδο και νομίζω ότι αυτό είναι άλλο ένα κίνητρο για τις ε, κυβερνήσεις για να συνεργαστούν ε, πιο άμεσα με την κοινωνία των πολιτών. Άλλο ένα παράδειγμα και τελειώνω. Όταν ήμουν στην Σλοβενία χρηματοδοτήσαμε ένα καταφύγιο για γυναίκες ε, που είχαν υποστεί εκμετάλλευση και υπεγράφει ένα μνημόνιο μεταξύ και, του κράτους Σλοβενίας και της ε, που το έκανε αυτό. Και είχαμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα το οποίο είχε τεράστιο αντίκτυπο στο τοπικό επίπεδο και μας δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η ε, βελτίωση που συχνά, της εμπιστοσύνης που συχνά δεν υπάρχει λόγω συγκρούσεων ή άλλων λόγων. Αυτή είναι η μεγάλη βελτίωση που πρέπει να επέλθει καθώς ε, πηγαίνουμε προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και μέρος της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Σχά και την κυρία Καλαβέρα και τον κύριο Φιουερέ. Δεν βλέπω άλλα μέλη να ζητούν το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συμμετέχοντες για τις συνεισφορές τους στην σημερινή συζήτηση και να θυμίσω ότι στην αρχή του επόμενου έτους η Επιτροπή μας ε, θα έχει μια συνάντηση με αντικείμενο της ενδιάμεσης επανεξέτασης και της δομής που θα ακολουθήσει μετά το 2020 και θα ήθελα να σας ξαναδώ όλους τώρα για να συνεχίσουμε τη σημερινή συνεδρίαση στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ όλους.